Euh, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, θα ομιλώ σιγά στην αρχή για να επιτρέψω σε όλους να πάρουν τις θέσεις τους. Χαίρομαι που ξεκινάμε με αυτή την σημαντική ακρόαση. Λέω εδώ για τους ομιλητές μας ότι δεν υπάρχουν και πολλοί στην αίθουσα. Υπάρχουν δύο βουλευτές, οι δύο πιο σημαντικοί για το απόγευμα. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται διαδικτυακά και το παρακολουθούν πολύ περισσότεροι εκτός εθούσης μεταξύ των οποίων και οι συνάδελφοι από τα γραφεία τους. Χαίρομαι που σας καλωσορίζω λοιπόν. Σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο θέματα τα οποία σε μια πρώτη φάση θα λέει κανείς δεν έχουν και πολύ σχέση μεταξύ τους. Απ' τη μία θα έχουμε ένα σημαντικό hearing για τα θέματα τα οποία έπονται του νομοθετικού πακέτου για την άμυνα εδώ και 5 χρόνια, 5-6 χρόνια. Μπορεί και 7. Και στο τέλος θα έχουμε λίγο χρόνο για ένα σημαντικό θέμα, την αξιολόγηση του κόστους της αμφισβήτησης των συμφωνιών του Σέγγεν. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για το πρώτο τμήμα τώρα, για την ουσία της απογευματινής συνεδρίασης. <coughs> Να υπενθυμίσω ποια είναι τα δεδομένα. Το 2009 πέρασαν δύο οδηγίες για την άμυνα. Η πρώτη αφορά τους ε, διαγωνισμούς και ε, δημόσιες αγορές. Και το δεύτερο, τη μεταφορά των αμυντικών προϊόντων ή των προϊόντων που σχετίζονται με την άμυνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει μια έκθεση εφαρμογής των οδηγιών αυτών μέχρι τέλος Ιουνίου. Η ακρόασή μας λοιπόν το απόγευμα σχετίζεται με την ουσία της υπόθεσης. Πρέπει να ακούσουμε κάποιες παρεμβάσεις που θα μας διαφωτίσουν σε σχέση με την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα επίσης να πω για όσους ε, θα πάρουν το λόγο και τους συναδέλφους που θα επωφεληθούν από τις σκέψεις σας ότι θα τεθούν ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο και κυρίως στην Επιτροπή. Να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν με ποιο λόγο θα είναι απαραίτητο να ξεκινήσει μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία μετά από την αναθεώρηση και αξιολόγηση της συγκεκριμένης οδηγίας σε λίγες εβδομάδες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος και αναφέρομαι στο παρελθόν. Το 2015 η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και η Πρόεδρος της είναι μαζί μας σήμερα έκανε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό και υπήρξε μια σημαντική συνεισφορά της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις δύο οδηγίες τις οποίες προαναφέρθηκα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε και την κυρία Γκάλπετ που είναι η συγγήτρια. Χαίρομαι που είναι μαζί μας η κυρία Γκάλπετς. Αυτά εισαγωγικά. Έχουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Σούμαν, και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο αμέσως στην πρόεδρο της Υποεπιτροπής Άμυνας και ε, Ασφάλειας, την κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ, πρόεδρε, συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν άκουσα την αγγλική διευμηνία. Δεν ήμουν εισηγήτρια της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας. Ήταν, ε, θα έλεγα, η έκθεση η οποία ξεκίνησε μετά από την πρωτοβουλία των συντονιστών της ΣΕΝΤΕ. Στα πλαίσια της αξιολόγησης λοιπόν της εφαρμογής των δύο αυτών οδηγιών, ασχοληθήκαμε με ένα πολύ σοβαρό θα έλεγα, καθοριστικό και ευαίσθητο πρόβλημα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε μία πρώτη φάση οι δαπάνες για την άμυνα αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των εθνικών προϋπολογισμών των χωρών μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν υποχρεώσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, υπάρχουν εθελοντικού τύπου συμμετοχές από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να φτάσουν στα α, όρια αυτά του 2% και ταυτόχρονα οι οδηγίες αυτές ψηφίστηκαν μετά από την αρχή μιας μεγάλης πολιτικής κρίσης και γι' αυτό όλοι πιστεύουμε ότι ο τομέας της άμυνας και η συνεργασία στον τομέα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το ε, μέγεθος των δημοσιονομικών ε, που αφιερώνονται στον τομέα αυτό και είναι μια ευκαιρία για την οικονομική ανάκαμψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ασφάλεια των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τους δύο αυτούς παράγοντες και να προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και στους δύο τομείς. Πρώτον, ευκαιρία ανάκαμψης μετά από οικονομική κρίση και από την άλλη να λάβουμε υπόψη μας τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καινούριε προκλήσεις, οι οποίες ε, μας βλέπουν να εξετάζουμε κάποια θέματα με καινούριο τρόπο. Η βασική δική μου δήλωση αφορά την σημερινή κατάσταση χωρών της δικής μου περιοχής. Μετά από την κομμουνιστική περίοδο στις χώρες μας εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη την σταθεροποίηση του αμυντικού τομέα για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε πλήρως και να επωφεληθούμε πλήρως από τα κοινοτικά μέτρα και στον τομέα της άμυνας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, λοιπόν. Περιμένουμε την αξιολόγηση του πακέτου συνολικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Σρίμαν, που είναι υποδιευθύντρια Γενική Υποδιευθύντρια στον τομέα της ανάπτυξης ε, και ασχολείται με την ε, υπόθεση στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ και θα ήθελα ε, να ε, συμφωνήσω με αυτά που μόλις υπόθηκαν ότι ε, στο πλαίσιο των σημαντικών απειλών κατά της ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να, να διατηρήσει μια ανταγωνιστική και καινοτόμα βιομηχανία άμυνας Θέλουμε λοιπόν να <clears throat> έχουμε ε, αμυντική βιομηχανία που να ε, ε, καλύπτει τις ανάγκες μας, αλλά και να έχουμε ισχυρή βιομηχανική βάση εντός της Ευρώπης. Οι δύο οδηγίες για τις συμβάσεις προμηθών στον τομέα της άμυνας και την απλούσευση των όρων και προϋποθέσεων της μεταφορές προϊόντων συνδεδομένων με τον τομέα της άμυνας είναι σημαντικές για την άμυνα στην Ευρώπη. Η πρώτη από τις οδηγίες Αυτέ αυτές ε, στόχο ε, έχουν να διασφαλίσουν τις διαδικασίες για τις διασυνορικές δημόσιες ε, συμβάσεις, αλλά να μπορούν και τα κράτη-μέλη να να προστατεύσουν τις, την άμυνα τους. Και η δεύτερη οδηγία έχει να κάνει με την καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την απλοποίηση των ε, κανόνων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεδομένων με τον τομέα της άμυνας. Έχουμε ένα νέο σύστημα αδειοδότησης. Αντί λοιπόν να ελέγχουμε εκ των προτέρων τις μεταφορές προϊόντων, ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη ε, να έχουν εκ των υστέρων ελέγχους για λιγότερο ευαίσθητα προϊόντα θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την αποτελεσματική εφαρμογή και των δύο οδηγιών και είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε αναλυτικά όταν υποβάλουμε την έκθεσή μας. Ε, καταλαβαίνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται τους στόχους αυτούς και χαιρόμαστε για τις θέσεις που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο επανειλημμένα. Πιο πρόσφατα, τον Μάιο του 2005, όσον αφορά τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης ε, και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση όσον αφορά τις δύο οδηγίες. Θα ξεκινήσω από αυτήν για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, όπως ε, είπατε και εσείς, αυτή τη στιγμή ε, αξιολογούμε την οδηγία αυτή. Η αξιολόγηση θα αποτελέσει τη βάση για την έκθεση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο που θα δημοσιευτεί αργότερα εντός της χρονιάς. Έχουμε όμως κάποια προκατακτικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση ε, στην ε, χρήση της οδηγίας αυτής, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Αυξάνεται η κοινοποίηση ε, σταθερά από 1.200 το 2012 σε πάνω από 3.000 κοινοποίησεις το 2015. Συνολικά είχαμε 9.000 από το 2011 μέχρι το 2015. Υπάρχει λοιπόν σαφής αύξηση αν κοιτάξουμε την αξία των συμβάσεων ε, υπό την οδηγία αυτή, βλέπουμε και εδώ ε, αύξηση από 1,5 ε, δισεκατομμύρια το 2012 μέχρι 30 δισεκατομμύρια το 2015 και πάλι πρόκειται για κάποια προκατακτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επαληθευτούν. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ε, κάποιες ε, σημαντικές ε, προμήθειες αμυντικού υλικού γίνονται εκτός του πλαισίου της οδηγίας και το παρακολουθούμε αυτό στενά. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση για να αποφύγουμε στρεβλώσεις στην αγορά. Επίσης είναι σημαντική η συνεργατική προσέγγιση μας. Προσπαθούμε να παρέχουμε προσανατολισμό και ολοκληρώνουμε τις ε, εργασίες ε, όσον αφορά ε, το, τους αποκλεισμούς κυβερνήσεων. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε τον στόχο ε, της πρόωθησης των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, κάτι που τονίστηκε και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου του 2015. Εργαζόμαστε πάνω στο πολύ σημαντικό αλλά δύσκολο αυτό θέμα στο πλαίσιο μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών αλλά και του σχετικού βιομηχανικού τομέα. Περιμένουμε να έχουμε τα συμπεράσματα της ομάδας αυτής το φθινόπωρο. Περνώ τώρα στο ε, δεύτερο μέρος της δέσμης μέτρων αυτών, που είναι η οδηγία για τις μεταφορές ε, προϊόντων. Ε, γίνεται αξιολόγηση που θα αποτελέσει τη βάση για την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του έτους από τις επαφές μας με τα κράτη-μέλη και τον βιομηχανικό τομέα ξέρουμε ότι τα νέα μέσα που προτείνονται στην οδηγία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως αναμενόταν. Υπάρχει λοιπόν ε, εδώ ε, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Γενικά οι άδειε ε, μεταφορών των κρατών μελών διαφέρουν πολύ όσον αφορά το περιεχόμενο, όσον αφορά δηλαδή το ποια προϊόντα καλύπτονται, αλλά και όσον αφορά τι προποθέσει. Υπάρχει λοιπόν σημαντικό κατακαιρματισμό στον τρόπο εφαρμογή τη οδηγία. Επίση, οι εταιρείε θα πρέπει να έχουν έγκριση για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις νέες άδειες. Ε, ε, όσο όμως ε, δεν υπάρχει πραγματική απλούστευση και έτσι προστιθέμενη αξία, θεωρούν ότι δεν αξίζει τον κόπο να προχωρήσουν στις διαδικασίες αυτές. Μέχρι στιγμής περίπου 40 επιχειρήσει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λάβει τη σχετική έγκριση, κάτι το οποίο ε, δεν ανταποκρίνεται στι προσδοκίε μα. Επίση, όσον αφορά την ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εναρμόνιση τη εφαρμογή ε, τη οδηγία για τι μεταφορέ προϊόντων Συνδεόμενων με, τον τομέα τη άμυνα, αυτά τα θέματα συμπεριλαμβάνουν έναν κατάλογο των μη ευαίσθητων προϊόντων και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την αδειοδότηση πιο ελκυστική για τις επιχειρήσεις. Ελπίζουμε ότι με την ε, συμμετοχική διαδικασία θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα όταν υποβάλουμε την έκθεσή μας σε εσάς όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Ε, τέλος, ε, κάτι στο οποίο νομίζω συμφωνούμε, πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερο όσον αφορά την εσωτερική αγορά στον τομέα της άμυνας εντός της χρονιάς. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει σχέδιο δράσης ε, για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και η αποτελεσματική εφαρμογή και των δύο οδηγιών θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του σχεδίου δράσης, αλλά πιστεύουμε ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να προχωράει πιο πέρα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ώστε να παράσχουμε κίνητρα ε, για καλύτερη αμυντική συνεργασία γενικά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, madame. Ε, Σας ευχαριστώ. και προφανώς και εμείς μοιραζόμαστε και έχουμε τους ίδιους ε, στόχους, το ξέρετε άλλωστε, για τις δύο αυτές οδηγίες. Προφανώς η αξιολόγηση που κάνετε για την εφαρμογή περιλαμβάνει διαφορετικά αποτελέσματα. Για τις μεταφορές προϊόντων θεωρείτε ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Αλλά θα τα ξαναδούμε αυτά όταν θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα περάσουμε λοιπόν στο πρώτο πάνελ. Να ευχαριστήσω όλους μας τους πανελίστες προσκεκλημένους που έχουν έλθει εδώ σήμερα το απόγευμα. Του εμπειρογνώμονές μα. Η πρώτη συζήτηση περιλαμβάνει δύο προσκεκλημένου. Και θα κοιτάξουμε λοιπόν την οδηγία για τι δημόσιε συμβάσει στον τομέα της άμυνας. Έχουμε δύο προσκεκλημένου. Ο δρ. Μάρτιν Τρίμπου, ο οποίος είναι καθηγητή ε, στην νομική σχολή του Birmingham και στη συνέχεια τον κύριο Τόμι Νόρτμπεργκ, ο οποίο είναι σύμβουλο ε, του Υπουργείου Άμυνα τη Φιλανδία. Δέκα λεπτά θα δώσω στον καθένα σα. Θα έχετε και διαφάνεια. Να χαμηλώσουμε ενδεχομένω και το φωτισμό για να φαίνονται καλύτερα οι διαφάνειε. Je vous donne la parole. allez Uh, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρωτού ξεκινήσω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που με προσκάλεσε. Ήμουν ο μοναδικός ακαδημαϊκός στο πάνελ και είναι μεγάλη τιμή και ευκαιρία για έναν ακαδημαϊκό να πάρει το λόγο εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρωτού ξεκινήσω να σας παρουσιάσω τα... την παρουσίασή μου το κατά πόσον ε, το εργαλείο της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας είναι αποτελεσματικό, ας θυμηθούμε καταρχάς ποιοι είναι οι στόχοι. Ο βασικός στόχος λοιπόν είναι να δώσει στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας ένα ειδικό, εξειδικευμένο εργαλείο προκειμένου η άμυνα και η ασφάλεια και ιδιαίτερως η εθνική ασφάλεια να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και στο στο εσωτερικό του μέσου αυτού και στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. Και άρα σκοπός είναι να μειωθεί η χρήση του άρθρου 346 της συνθήκης στην πράξη. Και αυτό γίνεται μέσω της χρήσης ε, της ε, οδηγίας 2004-18 για τις δημόσιες ε, υπηρεσίες ως το εργαλείο το οποίο θα δώσει μια εξειδικευμένη λύση στην οδηγία άμυνας και ασφάλειας χωρίς να χρησιμοποιεί το άρθρο 346. Αυτό το πετυχαίνει με τέσσερις τρόπους. Μέσω του περιορισμού, μέσω της ευελιξίας, μέσω της περιγραφής και μέσω της υποκατάστασης. Περιορισμός. Τι σημαίνει αυτό. Ότι έχουν προσταθεί αρκετές επιπρόσθετες εξαιρέσεις σε σχέση με το 2004-2018 που έχουν να κάνουν με την άμυνα σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ κυβερνήσεων, συνεργατικά έργα κτλ. κτλ. Ο τομέας λοιπόν, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής δεν είναι τόσο ευρύς όσο αυτός του δημοσίου τομέα. Ευελιξία, το βασικό κομμάτι, τι σημαίνει ότι δεν ε, ακολουθούμε πλέον την ανοιχτή διαδικασία που περιέχει το πιο πολύ ανταγωνισμό και περνάμε σε λιγότερο ανταγωνιστικές διαδικασίες, πιο πολύ μετά από διαπραγμάτευση. Άρα αυτή η οδηγία, σε αντίθεση με την οδηγία του δημοσίου κλάδου, επιτρέπει την ελεύθερη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πρώτερη ανακοίνωση του διαγωνισμού, με δηλαδή δημόσια σύμβαση και έτσι λοιπόν επιτρέπεται η μη χρήση ανταγωνισμού σε, σε πιο πολλούς τρόπους. Ο τελευταίος τρόπος που το προσαρμόζουμε αυτό στην ε, άμυνα είναι η υποκατάσταση. Η υποκατάσταση περιλαμβάνει και το δύσκολο ζήτημα των offsets, των αντισταθμισμάτων. Δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε αυτό το πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Εδώ θα προκαλέσω και θα πω κάτι ξεκάθαρα, γιατί τα αντισταθμίσματα είναι σχεδόν αδύνατο να συνδυαστούν και με την ιδέα με τη ελευθερή κυκλοφορία στην ιστορική αγορά και τη μη διακριτική μεταχείριση. Και είναι σημαντικό και αρνητικό στοιχείο ενδεχομένω για την νέα αγορά. Τι προβλέπει λοιπόν η οδηγία, δεν προβλέπει ξεκάθαρα αντισταθμίσματα. Ίσως ε, καλά κάνει, αλλά προτείνει κάτι εναλλακτικό το καθεστώ των υπεργαλαβιών. Και θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Τι λειτουργεί λοιπόν καλά και σωστά στην οδηγία αυτή και μετά στη συνέχεια θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Πολλά πηγαίνουν καλά γιατί πρόκειται για ένα καλογραμμένο νομοθέτημα το οποίο ε, πήρε μάλιστα χρόνια για την κατάρτισή του σε ό,τι αφορά την, το σκέλος του περιορισμού λειτουργεί από πολλές απόψεις και σε ένα βαθμό σε περιπτώσεις όπου θα χρησιμοποιούνταν το άρθρο 346 έχουν ε, πλέον μεταφερθεί σε αυτές τις ε, προβλεπόμενες εξαιρέσεις παρά το γεγονός ότι δεν ε, εξακολουθεί να πρόκειται για εξαιρέσει. Η ευελιξία του δυνατό σημείου τη οδηγίας και ιδιαίτερα η ελεύθερη χρήση της διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση του διαγωνισμού. Αυτό λειτουργεί πολύ καλά και θα πρέπει να συνεχιστεί έτσι ως βασική ιδέα. Η περιγραφή. Εδώ θέματα ασφάλειας ε, παροχής και προμήθειας περιγράφονται, επεξηγούνται στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ε, ανάθεσης και αυτό γίνεται σωστά και λαμβάνει υπόψη και το θέμα της ασφάλειας της πληροφορίας. Της πληροφορίας. Σε ό,τι αφορά το σύστημα τώρα ένωμων ε, μέσων, προστίθεται στην ε, οδηγία εκ των υστέρων. Δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προστασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό επιτυχές, παρά το γεγονός ότι είναι μάλλον ε, αρκετά κατακαιρματισμένα τα σχετικά στοιχεία που το υποδεικνύουν αυτό. Η οδηγία πλέον έχει εφαρμοστεί αν και καθυστερημένα σε όλα τα κράτη-μέλη και χρησιμοποιείται σε πολλά από αυτά τα κράτη-μέλη. Παρά το γεγονός ότι εδώ υπάρχει προφανώς μεγάλη ποικιλία. Κάποια κράτη-μέλη τα χρησιμοποιούν λες, και εδώ και πολλά χρόνια. Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα και κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα δημοσιεύσει ούτε ε, μία σύμβαση σχετική παρά το γεγονός ότι έχει πλέον ε, κλείσει, είναι πλέον ε, λειτουργική από το 2015. Άρα δηλαδή υπάρχει στη θεωρία αλλά δεν χρησιμοποιείται στην πράξη. Τι θα μπορούσε λοιπόν τώρα να βελτιωθεί, ας κοιτάξουμε. Χρειάζεται κάποια διευκρίνηση στο σημείο αυτό, ίσως ε, κάποιες προσθήκες, ίσως κάποιες διαγραφές σε κάποια σημεία. Και λίγο πιο πολύ υπόσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει σημειώματα καθοδηγητικών ε, στοιχείων για τις ε, κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά και τους νεοαποκτηθέντες εξοπλισμούς και η εξαίρεση για τους διεθνείς οργανισμούς θα πρέπει να διευκρινιστεί, αλλά αυτό έχει δρομολογηθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογής, αναρωτιέμαι κατά πόσον θα μπορούσε να υποβληθεί η οδηγία από το προσάρτημά της, ε, παρεθμώντας κατά μη εξαλειπτικό τρόπο τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κάποιοι εμπειρογνώμονε. μας αναφέρουν ότι ο τρόπος που περιλαμβάνεται τώρα είναι μάλλον, προκαλεί μάλλον σύγχυση σε ό,τι αφορά την διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η πρόβλεψη της οδηγίας, αν και δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται ένας διάλογος, ανταγωνισμό, όταν επιτρέπεται την ελεύθερη χρήση της διαδικασία διαπραγματεύση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της, ε, του διαγωνισμού. Φυσικά αυτό αποτελεί μια κατευθυντήρια γραμμή, αν και πολύ λίγες ε, χώρες ε, χρησιμοποιούσαν τον διάλογο τη συζήτηση αυτή για τις διαπραγματεύσεις, πόσο μάλλον στο, σημείο στον κλάδο της άμυνας τα αξιοποιούσαν αυτά. Το με το Βασίλειο. Ίσως λοιπόν αυτός ο διάλογος περί ανταγωνιστικότητας θα μπορούσε να διαγραφεί καθώς επιτρέπεται αυτή η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Από την άλλη πλευρά, η ανοιχτή διαδικασία δεν συμπεριλαμβάνεται στο μέσο αυτό και υπάρχουν κλάδοι όπου χρησιμοποιείται αυτό θα πυρομαχικά σε κάποιε περιπτώσει της συντήρηση και ενδεχομένω εκεί θα έπρεπε να α, χρησιμοποιείται όχι υποχρεωτικά, αλλά να επιτρέπεται αυτή η ελεύθερη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Αναρωτιέμαι δηλαδή, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις σαν αυτές δεν ε, συμπεριλαμβάνεται ως δυνατότητα. Κάτι άλλο που μας συνδέει με το επόμενο θέμα στην οδηγία ICT. Το θέμα της ασφάλειας της προμήθειας, του ανεφοδιασμού είναι σημαντικό στην οδηγία και νομίζω ότι όταν ο αγοραστής είναι Υπουργείο Άμυνας άλλου κράτους, γιατί θα πρέπει αυτό να υπόκειται σε οποιαδήποτε υποχρέωση αντιδότησης. Ούτε τα Υπουργεία Αμήνης δεν μπορούμε να, να εμπιστευτούμε των 28 κρατών μελών. Δεν θα ήταν λοιπόν μια ιδέα να εξαιρεθούν τα Υπουργεία Άμυνα ως αγοραστές από την ε, οποιαδήποτε επιβολή υποχρέωσης αντιοδότησης να υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Αυτό γίνεται με την οδηγία όσο έχει και ενδεχομένω να μην χρειάζεται και αλλαγή της οδηγίας. γιατί αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά με θέματα εφαρμογή. Μία ιδέα αναφέρω μόνο και για τα αντισταθμίσματα, τι αντισταθμίσει. Οι κανόνε υποκατάσταση είναι πολύ περίπλοκοι. Κανεί δεν του χρησιμοποιεί, όλοι του φοβούνται. Αλλά, και εδώ θα κλείσω, νομίζω ότι είμαστε αρκετά. Βιαστήκαμε αρκετά γιατί θεωρούσαμε ότι το 2016 όλοι θα είχαν εφαρμόσει την οδηγία από το 2011 και θα είχαμε ήδη μία πενταετή εμπειρία. Όμως αυτό δεν έγινε. Χρειάζεται πιο πολύς χρόνο γιατί άργησε και η μεταφορά και η εφαρμογή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μας είχατε πει ότι αυτό το οποίο απαιτείται για την άμυνα είναι ειδικά μέτρα. Και τα ειδικά αυτά μέτρα και σταθμά πρέπει να εφαρμοστούν και στα πλαίσια των οικονομικών προβλέψεων. Και υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς βέβαια, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Φώτιγκα. Περνάω στον δεύτερο μιλητή, ο κύριος Νόρμπεργκ. Εσείς είστε από την άλλη πλευρά κατά κάποιο τρόπο κύριε Τόμι Νόρντμπεργκ. Είστε ο πελάτης αν θέλετε, είστε ο χρήστης αυτής της οδηγίας, είστε ο οργανωτής. Βρίσκεστε σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πρακτικά θέματα σε σχέση με τη συγκεκριμένη οδηγία. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε σήμερα να έρθω εδώ να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω, όπως υπόθηκε, τη θέση ενός μικρότερου κράτους μέλους. Uh, I will use the opportunity to... Θα αδράξω την ευκαιρία να πω λίγα λόγια για τη Φιλανδία και το σύστημά μας για να αποκτήσετε μια ιδέα του από πού ε, ερχόμαστε ως αγοραστής ε, στην αγορά ε, αμυντικών προϊόντων της Ευρώπης. Η Φιλανδία δεν έχει συμμάχους, είναι ουδέτερη χώρα. Όπως βλέπετε έχουμε χερσαία σύνορα σημαντικού μήκους με την Ρωσία. Επίσης έχουμε ακόμα Έχουμε ακόμα στρατιωτική θητεία. Όλοι οι άντρες ε, λοιπόν ε, κανονικά περνούν στρατιωτική θητεία και δίνουμε μεγάλη σημασία στην ε, ασφάλεια προμηθειών λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και επειδή είμαστε ουδέτερη χώρα, ο προϋπολογισμός μας στην άμυνα ανέρχεται περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και περίπου 600.000 ευρώ επενδύουμε. Υπάρχουν ε, ε, ανά έτος, αλλά αυτές είναι σε γενικές γραμμές Αυτά είναι σε γενικέ γραμμέ τα ποσά. Γενικά, ο σχετικό ε, τομέα μα κυριαρχείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σημαντικό για μας είναι ότι θεωρούμε ότι η σχετική βιομηχανία στη χώρα μας αποτελεί ε, αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας άμυνας. Ο σχετικός τομέας μας εξάγει το 40 με 60% των προϊόντων του. Επειδή λοιπόν η εγχώρια αγορά δεν είναι μαζική, είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις μας ε, να εξάγουν και προϊόντα εκτός των συνόρων μας. The European Έχουμε πενταετή πείρα με την οδηγία και φαίνεται να υπάρχει ακόμα ισχυρή προτίμηση για εθνικές ε, αγορές και νομίζω ότι και η αξιολόγηση της Κομισιόν ε, το δείχνει αυτό. Και γενικά η αλυσίδα τροφοδότησης ε, ακολουθεί εθνικές γραμμές και υπάρχει έλλειψη ε, ε, διεθνούς συνεργασίας. Επειδή είμαστε μικρό κράτος μέλος, επειδή είμαστε χώρα αγοραστής περισσότερο, πράγμα που σημαίνει ότι λόγω στην περιορισμένη βιομηχανική βάση μας δεν μπορούμε να βρούμε όλα τα αμυντικά συστήματα που θέλουμε στην πατρίδα μας. Πρέπει να προσφεύγουμε και στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές χώρες και σε τρίτες χώρες για τις αγορές μας. Τι ψάχνουμε λοιπόν. Καταρχάς ε, θέλουμε κατάλληλο εξοπλισμό για τις ε, ε, στρατιωτικές δυνάμεις μας. Χρειαζόμαστε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε να εκτελούμε τις αποστολές μας και εντός της χώρας και να ανταποκρινόμαστε στα διεθνή καθήκοντά μας. Και αυτό που αναζητούμε είναι αξία σωστή σε σχέση με τις δαπάνες μας. Σε καιρούς ε, οικονομικής κρίσης έχουμε και εμείς περικοπές στον προϋπολογισμό μας. Γι' αυτό η ε, κυβέρνηση της ε, Φιλανδίας αναμένει το Υπουργείο Αμήνης να κάνει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες αγορές. Όσον αφορά τον σχετικό τομέα και την αγορά, στόχος μας είναι να έχουμε ανταγωνιστική βιομηχανική βάση σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό για μας, διότι όπως σας είπα νωρίτερα, θεωρούμε την αμυντική βιομηχανία τομέα ζωτικής σημασίας για την προστασία ε, των ε, συμφερόντων μας και της ασφάλειας μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα νέα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ναι πράγματι, αποτελούν εργαλεία της εσωτερικής αγοράς, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ωστόσο, τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά την αξιολόγηση και την πιθανή τροποποίηση της οδηγίας ή κατά τη διαμόρφωση νέων πολιτικών. Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Καταρχάς πιστεύουμε ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η κοινή κατανόηση των προβλημάτων. Έχουμε τις μεγάλες χώρες παραγωγούς και τις μικρότερες χώρες αγοραστές που έχουν τον δικό τους αμυντικό τομέα, αλλά δεν νομίζω ότι βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Και χρειαζόμαστε όχι μόνο κοινή κατανόηση του προβλήματος, αλλά και ε, κοινή θέση όσον αφορά τις πιθανές λύσεις και πέρα από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επίσης είναι σημαντικός ε, ενδιαφερομένος, αλλά μιλάμε και για τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθούν κίνητρα. Να δημιουργηθούν κίνητρα ε, για μια αγορά με περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία κατά την ε, δημιουργία κινήτρων θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη αγορά. Ουσιαστικά δεσπόζεται από τις κυβερνήσεις ένας πελάτης υπάρχει στην ουσία. Πρέπει όμως ε, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου να υπάρχουν ε, κίνητρα για τους μεγάλους προμηθευτές να είναι ανοιχτή απέναντι στο σύνολο της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει να εξαλείψουμε τα εμπόδια θα πρέπει να εξαλείψουμε εμπόδια που αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, στην διασυνοριακή συνεργασία και μεταξύ κρατών μελών, αλλά πιθανότατα και, ανάμες και εντός του βιομηχανικού τομέα. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε αλυσίδια προμηθειών που να συμπεριλαμβάνει προμηθευτές από μεγάλες και μικρές χώρες ώστε να εκμεταλλευτούμε ε, τα μέγιστα την δυνατότητα καινοτομίας που υπάρχει στον τομέα αυτών. Merci beaucoup, Monsieur Nordberg. Vous nous avez dit souvent que vous étiez issu d'un pays que vous considériez comme un petit pays de l'Union. C'est vous εσείς ε, είπατε ότι είστε μικρή ε, χώρα ευρωπαϊκή και ακόμα και σε μια χώρα που δεν είναι από τις μεγαλύτερες, η άμυνα ανεξαρτήτως του μεγέθους είναι μια μεγάλη υπόθεση. Μας είπατε ότι βρίσκεστε σε μια φάση εθνικής ολοκλήρωσης. Ε, θα συμφωνήσω με την τελευταία σας διαφάνεια Πράγματι οι στόχοι τους οποίους θέσατε είναι κοινοί. Μας είπατε παράλληλα ότι απαιτείται χρόνος, ότι στην ουσία η χώρα σας ξεκινά στην διαδικασία ε, τώρα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκαλπέλτς, η οποία είναι συνεισηγήτρια από το 2015 σε σχέση με τις ε, δύο παρεμβάσεις οι οποίες προηγήθηκαν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και φιλοξενούμενοι, σας ευχαριστώ για ε, την παρέμβαση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πιστεύουμε ότι η αγορά της άμυνας είναι μια πολύ ειδική ε, μορφή αγοράς οι παραδοσιακές αντιλήψεις για την ελεύθερη αγορά δεν λειτουργούν πλήρως εδώ και γι' αυτό αυτό το οποίο θα θέλαμε να πετύχουμε είναι να καταστεί η αγορά αυτή ανταγωνιστική. Χαίρομαι λοιπόν βλέποντας ότι η συγκεκριμένη οδηγία έχει αρχίσει και εφαρμόζεται με επιτυχία αν και βέβαια δεν θα διαφωνήσω με αυτό το οποίο ακούστηκε, ότι ναι μεν έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά παραμένει ιδιαιτέρως ε, πολυδιασπασμένη. Δεν έχουμε από την άλλη ανάγκη για υπερβολικές παρεμβάσεις στην αγορά αυτή και θα συμφωνήσω με τον ομιλητή ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι να επιτρέπουν τις ελεύθερες επιλογές, θα έλεγα, στον τομέα των προμηθειών αμυντικού υλικού. Και θα πρέπει να αφήσουμε ε, τους ε, εμπλεκόμενους σε κάθε χώρα να κάνουν τις σωστές επιλογές οι υπερβολικές ρυθμίσεις και διακανονισμοί εμπλέκουν τα πράγματα. Είναι πάντως απαραίτητο η εσωτερική αγορά να είναι ελεύθερη εμποδίων και θα πρέπει να κάνουμε βήματα τουλάχιστον για να μειώσουμε τα συγκεκριμένα εμπόδια. Όταν διατύπωσα την έκθεση αυτή είχαν ήδη τεθεί αρκετές ερωτήσεις και είχαν γίνει ζωηρότατες συζητήσεις μεταξύ των οποίων ε, τίθεται και το θέμα των αντισταθμισμάτων, των αντισταθμιστικών μέτρων. Και εδώ θα συμφωνήσω λίγο με αυτά τα οποία είπε ο ένας από τους ομιλητές για τα αντισταθμιστικά αλλά να πω επίσης ότι πολλές φορές τα αντισταθμιστικά αντί να λειτουργήσουν θετικά λειτουργούν αρνητικά για την πλήρη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα θέλαμε επίσης στο μέλλον μετά από την ενδιάμεση αναθεώρηση να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί σαν μια πραγματική ενιαία αγορά. Γιατί όπως είπε ο κύριος Νόρμπερκ, Κάποιες χώρες ε, και μικρές και μεγάλες και δεν αναφέρομαι μόνο στη Φιλανδία λειτουργούν με πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Οι πολιτικές ε, ε, μπορεί να είναι κοινέ εφόσον η κοινή πολιτική είναι κατάλληλη για το σύνολο των χωρών. Απαιτείται λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή να γίνουν περισσότερα βήματα. και οι κυρώσεις αν χρειαστεί μπορεί να οδηγήσουν σε βελτιώσεις. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν επίσης κίνητρα. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν στοιχεία ενθάρρυνσης για την περαιτέρω ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ε, είναι μια σημαντική ενημέρωση που θα χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη εκθεσή μας. Ε, ευχαριστώ ε, ήρθε ο κύριος Σβάμπο, εισηγητής, ο συντονιστής μάλλον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν ξέρω, Ανδρέας, αν θες να κάνεις κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και καταρχάς χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα το απόγευμα ασχολούμαστε με το σημαντικό αυτό θέμα για την εσωτερική αγορά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να του συγκεκριμένου μας και να τους πω ξεκάθαρα ότι και εμείς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα καθημέλη πάντα στο θέμα των ε, προϊόντων αμήνη. αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει υπερβολική προσέγγιση, υπερβολική επικέντρωση στη επίπεδο της ε, εθνικών κρατών μελών και πριν από κάποιε εβδομάδες ψηφίσαμε την οδηγία την NIS για τα ζητήματα αυτά και μας χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος γιατί ε, ακόμα και σε αυτή την ψηφιακή εποχή το θέμα ε, της εθνικής ασφάλειας έχει αλλάξει περιορισμένα μόνο. Και φυσικά υπάρχει το θέμα της κυριαρχίας αλλά σε ό,τι αφορά την συνοριακή ασφάλεια των ε, ψηφιακών υπηρεσιών υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διασύνδεση των ε, εθνικών συστημάτων ασφαλείας και θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και από κοινού να οργανωθούμε και νομίζω ότι αυτό που φάνηκε και από τις παρουσιάσεις είναι ότι δεν έχουμε προχωρήσει επαρκώς στον τομέα της άμυνας προς την κατεύθυνση αυτή και όπως είπε και η κυρία Γκάλ Η Επιτροπή ΙΜΚΟ πάντα επισημαίνει και το άρθρο 96 της συνθήκης για να μην υπάρχει υπερβολική επικέντρωση στα εθνικά κριτήρια και γι' αυτό λοιπόν προσβλέπω και στο δεύτερο ήμιση της σημερινής ακρόασης για να δούμε ποιο θα είναι τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα πρότεινα αν θέλετε να πάρουν το λόγο οι δύο από ένα λεπτό ο καθένας αν θέλουν να απαντήσουν στα θέματα που, που έθεσαν οι ίδιοι ή στα θέματα που έθεσαν οι ευρωβουλευτές. Κύριε Τριμπούς, θα θέλετε να πάρετε το λόγο για να κάνετε κάποια παρατήρηση ενδεχομένω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα θέμα το οποίο ήθελα να δείξω σε ό,τι αφορά ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πρώτης παρουσίασης είναι το εξής, ότι Αντί να υπάρχουν κυρώσεις, θα έπρεπε να υπάρχουν μάλλον κίνητρα. Η οδηγία κινείται πιο πολύ στη γραμμή των κυρώσεων. Αυτό δεν έχει ακόμα αποκρισταλωθεί. Η πίεση δεν θα προέλθει πιο πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εξαναγκάσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις διτάξεις της οδηγίας. Η πραγματική α, πίεση θα είναι για τα εθνικά δικαστηρία όταν οι υποβάλλοντες ε, προσφορές που θα έχουν ε, θα υποβάλουν καταγγελίες και θα χρησιμοποιήσουν το δικαστικό σύστημα για να ανασταλούν οι διαδικασίες, να ξαναπροκηρυχθεί διαγωνισμός. Εκεί θα είναι η πραγματική πίεση. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Δεύτερη παρατήρηση. Πολύ χαίρομαι που επιτέλου κάποιος το λέει αυτό γιατί δεν τονίζεται επαρκώς. Ότι δίδεται πάρα πολύ έμφαση στο θέμα της εθνικής ασφάλειας. Και δεν αντιλέγω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αντεπιχείρημα κατά της ενιαίας αγοράς. Αν το αντιληφθούμε αυτό ότι σε ό,τι αφορά τη συνθήκη και την οδηγία πάντα υπάρχει αυτός ο ελοχεύων κίνδυνος να καταλήξουμε σε κατάχρηση και το περιγράφουμε ως εθνική ασφάλεια, αλλά ουσιαστικά δεν πρόκειται για εθνική ασφάλεια. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε λοιπόν να πατάξουμε τον κίνδυνο αυτό, πολλά θα έχουμε κερδίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριο Νόρμπεργκ. Αν θα θέλει να πάρετε το λόγο να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και θα ήθελα να σχολιάσω καταρχά αυτά που είπε, αυτά που ακούσαμε για ανάγκη μεγαλύτερη συνεργασίας για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Νομίζω ότι τα δύο αυτά ζητήματα μπορούν να συνδυαστούν. Δεν αποκλείει το μέντο δε. Από πλευράς κυβέρνησης πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς ε, της άμυνας που προορίζονται μόνο για εθνική χρήση, αν θέλετε. Αυτό είναι διαφορετικό ανά χώρα, αλλά πάντα υπάρχουν τέτοιοι τομείς και πάντα δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι είναι εκτός του πεδίου αυτού αποκλειστική εθνική ε, χρήση. Ε, σε αυτού του τομεί θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων. Ένα παράδειγμα να σα δώσω. Πριν από κάποια χρόνια η Φιλανδία εξέταζε ε, ψάχνει μάλλον μεταλλικές δεξάμενες γιατί θέλαμε να αυξήσουμε τον εξοπλισμό μας και μπορούσαμε λοιπόν τότε είτε να αυξήσουμε ε, τις, πρώτη, τις εγκαταστάσεις που είχαμε ή να πάμε στην αγορά και να αγοράσουμε ναι, σε τέτοιες δεξαμενές ή να αγοράσουμε τρίτη λύση πλεονασματικά τέτοια προϊόντα από μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό ήταν πραγματικά η κατά πολύ πιο συμφέρουσα λύση. Και αυτοί ξεφορτώθηκαν το πλεόνασμα και βγάλαν κάποια χρήματα και εμείς είχαμε την καλύτερη τιμή. Και αυτή λοιπόν η δραστηριότητα, αυτή η αγοραπολισία έγινε εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα παράδειγμα ενό ιδιαίτερου χαρακτηριστικού και είναι παράδειγμα, αν θέλετε, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Άρα, ναι, μεν πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν ευαίσθητα εθνικά συμφέροντα για την εθνική ασφάλεια, αλλά πέρα από αυτά υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο περιθώριο συνεργασία και πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωση τη λειτουργία τη αγορά μα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αυτό που λέτε είναι σχεδόν διασκεδαστικό. Βέβαια είναι κυρίως ενδιαφέρον. Μιλάμε πολλές φορές για την αναδιαναμητική οικονομία, για την κυκλική οικονομία ε, και εδώ τίθεται το θέμα της συνεργασίας των κρατών μελών και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί ότι ακόμα και σε αυτό τον τομέα η, η οικονομία αυτή η συνεταιριστική παίζει κάποιο ρόλο. Κύριε Τρίμπους, σωστά μιλήσατε και για τις κυρώσεις, όχι τόσο τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί άλλο είναι να αποφασίζει κανείς, άλλο να τις εφαρμόζει. Αλλά για το δικαστικό επίπεδο και για το σύνολο των κρατών μελών, Μία από τις βασικές θα έλεγα θετικές πλευρές είναι το να παίρνει κανείς αποφάσεις, αλλά δεν θα πρέπει οι αποφάσεις αυτές να είναι λανθασμένες σε τόσο στρατηγικούς τομείς. Έχετε δίκιο λοιπόν. Να περάσουμε τώρα σας παρακαλώ στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για την οδηγία. Έχουμε δύο εμπειρογνώμονες. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Καρλιέ, ο οποίος είναι υπεύθυνος στην Γενική Γραμματεία Άμυνας και Ασφάλειας για τα θέματα των προμηθειών εκεί όπου αποφασίζονται εν πάση περιπτώσει τα πράγματα και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Τσίλβερς ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά στη Rolls Royce. Κυρία Καγλίε, έχετε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και από γαλλική πλευρά να κάνω έναν μικρό απολογισμό για τον τρόπο που εφαρμόζουμε την οδηγία και πόσο συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως το θυμήσατε, για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε πιο εύκολα τα μέσα που παρέχει η οδηγία και πώς θα συνεχίσουμε να την εφαρμόζουμε σωστά και να εναρμονίσουμε καλύτερα τις διαδικασίες. Εξ θα ήθελα να πω ότι στη Γαλλία θεωρήσαμε ότι η οδηγία αυτή είναι το καθοριστικό κομμάτι αν θέλετε το οποίο πρέπει να ε, εφαρμοστεί για την καλύτερη εδραίωση και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ε, βιομηχανίας της άμυνας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε το supply chain ε, των αμυντικών μας βιομηχανιών, οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερο διεθνείς. Θα πρέπει λοιπόν να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι το 2010 και τα οποία βάριναν τις βιομηχανίες μας σε διοικητικό και διακανονιστικό επίπεδο και δεν τους έδιναν την δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επρόκειτο για, ένα βασικό, για μια βασική τροχοπέδη ε, στην ανάπτυξη της τεχνολογικής αμυντικής μας βάσης. Οι κοινοτικέ ρυθμίσεις έχουν ακριβώς σαν στόχο να βελτιώσουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Στη Γαλλία κάναμε δύο πράγματα. Από τη μία προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε με τον πλέον ορθό τρόπο την συγκεκριμένη οδηγία από το 12 και μετά, την εγγράψαμε στο εθνικό δίκαιο και ταυτόχρονα με την ευκαιρία αυτή αναθεωρήσαμε το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών αμυντικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αλλά παρόλα αυτά μπορέσαμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε την μεταρρύθμιση σε βάθος του συστήματός μας. Ε, στο παρελθόν για την εξαγωγή πολιτικού υλικού είχαμε το σύστημα προκαταρκτικής έγκρισης και μετά αδειοδότησης εξαγωγής. Ενώ τώρα ενιοποιούμε τα δύο αυτά συστήματα Κάτι το οποίο επιτρέπει στους ε, εκπροσώπους της βιομηχανίας να απλοποιήσουν τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα δημοσιεύσαμε ε, δέκα διαφορετικές τέτοιου τύπου άδειες και ε, ενεγράφησαν δέκα αμυντικές βιομηχανίες από τις 48 όπως υπενθύμισε η Επιτροπή. Η πιστοποίηση είναι το μέσο που επιτρέπει για ένα σύνολο βιομηχανιών ή για την υπεύθυνη για ένα πρόγραμμα επιχείρηση να μπορεί να προμηθεύεται υλικά χωρίς να ζητά κάθε φορά ειδική αδειοδότηση για μια ολόκληρη σειρά υλικού από υπεργολάβους παροχής προϊόντων που είναι σε άλλες χώρες της αλυσίδας προμηθειών και εφόσον είναι προεγγεγραμμένες και προπιστοποιημένες έχουν την δυνατότητα να εισάγουν τα προϊόντα και να τα επανεξάγουν μετά στο σύνολο ε, της ε, δραστηριότητάς τους. Υπόθηκε ήδη και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τώρα μετά από μία πρώτη περίοδο της οδηγίας είναι ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα Όλοι έχουμε ευθύνες και το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι η οδηγία μας δίδει πράγματι όλα τα μέσα τα οποία έχουμε ανάγκη, μέσα τα οποία είναι ισχύρα και τα οποία όμως δυστυχώς υποχρησιμοποιούνται στην παρούσα φάση γιατί ελείπουν τα στοιχεία συντονισμού. Όλα τα κράτη-μέλη δεν πόρεσαν να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία με την ίδια ταχύτητα και να τα μεταφέρουν ε, στα εθνικά του συστήματα. Αυτό εξηγείται βέβαια. Όταν μιλούσαμε στο παρελθόν για τα διοικητικά εμπόδια, ξέρουμε ότι είχαμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Πάντως προσπαθήσαμε σε μία πρώτη φάση να ε, ε, συνεργαστούμε με τις χώρες του πλαισίου δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Γαλλία και Γερμανία και να κάνουμε κάποιες προτάσεις ε, συνολικές με τις οποίες ε, φτάσαμε στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είναι μια μέθοδος η οποία λειτουργεί αρκετά καλά. Το κάναμε αυτό μέσα από μια πρώτη φάση τον Ιανουάριο του 2015, όπως είπε πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν να ενισχύσουμε την χρήση των γενικών αδειοδοτήσεων εναρμονίζοντας ε, τις διαδικασίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κάναμε ε, προτάσεις για δύο γενικές αδειοδοτήσεις. Η μία αφορά τις ένοπλες δυνάμεις των 28 χωρών και η άλλη αφορά ακριβώς τις πιστοποιημένες βιομηχανίες, διότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα της οδηγίας Στη συνέχεια μας φάνηκε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να βελτιώνουμε τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη, εναρμόνιση των καταλόγων προϊόντων και να καταστήσουμε πιο ελκυστικά τα μέσα της οδηγίας, όπως την πιστοποίηση και τις γενικές άδειες. Ένα τελευταίο στοιχείο ίσως λίγο τεχνικό. Εδώ ο εκπρόσωπος της SDE θα επανέλθει. Οι βιομηχανοί έχουν την ανάγκη μια μέθοδο που να επιτρέπει την ταξινόμηση του στρατιωτικού υλικού. Αν εγώ είμαι βιομήχανος και σχεδιάζω ένα υλικό, αν θα είναι αποκλειστικά στρατιωτικής χρήσης ή θα είναι προσαρμοσμένες για τη λεγόμενη διτή ή διπλή χρήση. Ε, και το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και εδώ ακριβώς τίθεται το θέμα των, της φραγίδας, αν θέλετε, της σήμανσης που λέει ότι ε, υλικό σχεδιασμένο για στοχιωτική χρήση. Συνεχίζουμε από το 2015 λοιπόν την ανάλυση της κατάστασης ε, με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά έτσι ώστε να καθοδηγήσει ε, τις προσπάθειες αυτές. Έχουν δημιουργηθεί Οκτώ ομάδες εργασίας έχουν συνεδριάσει, μάλλον οκτώ ομάδες, επτά ομάδες εργασίας από το 2014 και μετά. Και τον τελευταίο χρόνο καταφέραμε να εναρμονίσουμε ένα πρώτο κατάλογο υλικού γνωστού στα κράτη-μέλη. Αυτό μας έλειπε στο παρελθόν. Για δύο λοιπόν γενικές άδειες προς τις ένοπλες δυνάμεις από τη μία και τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις από την άλλη. Το δεύτερο θέμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και εδώ ε, τα αρχικά κρατημέλη έκαναν κάποιες πρώτες προτάσεις πάνω στις οποίες ε, συζητάμε με τις 22 υπόλοιπες χώρες και την Επιτροπή είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει με, τα, ε, ε, με τις επανεξαγωγές προς τις χώρες της Ένωση. Δεν αρκεί να εναρμονίζουμε την κυκλοφορία των προϊόντων σε μία πρώτη φάση στο εσωτερικό, αλλά και προς τρίτες χώρες. Και εδώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις πρακτικές που ακολουθούνται στις διάφορες χώρες. Αυτή είναι η προσπάθεια στην παρούσα φάση. Ε, έχουμε ένα κατάλογο υλικού για τις πιστοποιημένες βιομηχανίες και για τις ένοπλες δυνάμεις. Εναρμονίζουμε τις συνθήκες επανεξαγωγής και ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια κλειστή λίστα, ένα κλειστό κατάλογο χωρών εμπιστοσύνης εκτός της Ένωσης, όπου θα μπορούμε να εξάγουμε το σύνολο των προϊόντων, τα οποία εντάσσονται στις δύο ε, συνολικές ρυθμίσεις που ανέφερα προηγουμένως, στις δύο συνολικές άδειες. Επίσης, ε, εμβαθύνουμε την σήμανσή μας αυτή στην οποία αναφέρθηκα, το ειδική σχεδίαση για στρατιωτική κρίση. Εδώ υπάρχει εφέρον από τις στρατιωτικές βιομηχανίες και έχουμε και καλό input από τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες στα πλαίσια της αναθεώρησης των προϊόντων των υλικών των στρατιωτικών προς εξαγωγή έχουν την ίδια προβληματική. Οι προσπάθειες που κάνουν οι Αμερικανοί φυσικά και αυτή ε, ε, η προσπάθεια μάλλον έχει σαν στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Αμερικανικής βιομηχανίας. Θέλουμε να καταστήσουμε τη διαδικασία πιστοποίησης ελκυστική και θέλουμε να απλοποιήσουμε την διαδικασία αυτή πιστοποίησης, η οποία μέχρι τώρα θεωρείται ότι ήταν μακρόχρονη και κοστοφόρα, ενώ τώρα προσπαθούμε να, ε, ε, την, να βελτιώσουμε τις δύο αυτές συνθήκες. Συμπερασματικά, βλέπετε ότι εμείς στην Γαλλία θεωρούμε ότι τα μέσα της οδηγίας είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την ανέρεση των, εμποδίων στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής αλυσίδας προμηθειών. Αυτό το οποίο συνεχίζει να ελείπει όμως είναι η πλήρης εναρμόνιση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και αυτό το οποίο λείπει είναι η καλύτερη χρήση από ό,τι σήμερα αυτών των υλικών. Έχει υπάρξει πρόοδος εδώ και δύο χρόνια στο εσωτερικό της Ένωσης, μένει όμως να γίνουν πολλά αυτή στιγμή ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες αυτές, τότε θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε πραγματικά από την συγκεκριμένη οδηγία. Άλλωστε θεωρούμε ότι το Συμβούλιο του 2016, τον Ιούνιο του 2016, όταν θα γίνει και η πλήρης διαμόρφωση του σχεδίου δράσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τις ωφέλειες που μπορούμε να βγάλουμε από την οδηγία. Euh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρλιέ. Ο επόμενο ομιλητής ενδεχομένω να απαντήσει εν μέρη και σε αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά την αντίδραση των επιχειρήσεων και ενδεχομένω να μην υπάρχει η ίδια στάση από πλευρά των επιχειρήσεων. Να δώσω λοιπόν το λόγο πάρα αυτά στον κύριο Σπένσερ Τσόιλβερ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα. Ε, εκπροσωπώ την ε, Ένωση ε, βιομηχανιών ε, της άμυνας ε, και του διαστήματος. Δεν εκπροσωπώ λοιπόν τη Rolls Royce σήμερα. Τέσσερις τομείς θα ήθελα να εξετάσω σήμερα. Την εφαρμογή της οδηγίας μέχρι τώρα, τις αδυναμίες, τις θετικές εξελίξεις και το τι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Καταρχάς όσον αφορά την εφαρμογή. Νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ήταν αργή η πρόοδος και υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Καταρχάς, ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη εξετάζουν τις μεταφορές προϊόντων κατά περίπτωση και εκδίδουν ε, ξεχωριστές ε, άδειες για συγκεκριμένες μεταφορές, ενώ δεν χρησιμοποιούν γενικές άδειες που επιτρέπουν πολλαπλές μεταφορές προϊόντων. Και γι' αυτό καθυστέρησαν αρκετά μέχρι να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτές τις γενικές άδειες και να βρουν τους νέους τρόπους εργασίας. Επίσης, ε, σημαντικός, ε, τομέα, ε, σημαντικός λόγος για την καθυστέρηση ήταν η έλλειψη καθοδήγησης. Κάποια κράτη-μέλη έχουν εκδώσει σχετική νομοθεσία, πιο αναλυτικές καθοδηγητήριες γραμμές όμως έχουν εκδώσει πολύ λίγα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, βασικό καινοτόμο στοιχείο της οδηγία ε, ήταν η πιστοποιημένη εταιρεία, η οποία ε, στόχο είχε να είναι μέτρο οικοδόμησης της εμπιστοσύνη. Στην αγορά ήθελαν να έχουν την εγγύηση ότι το κράτος μέλος που θα λαμβάνει κάποιο υλικό μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις οδηγίες. Αλλά λίγα προγράμματα συμμόρφωσης εταιριών υπήρχαν και έτσι ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί το καθεστώς ε, των εταιριών. Γι' αυτό ε, κάποια κράτη-μέλη έπρεπε να ε, δημιουργήσουν σχετικά συστήματα, κάτι που απέτυχε αρκετό χρόνο. Επίσης, σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή της οδηγίας μέχρι τώρα ήταν η ασάφεια όσον αφορά τις γενικές άδειες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. ενώ ήταν σαφές βήμα προόδου το θέμα της βάσης δεδομένων των κρατών μελών, οι άδειε που έχουν εκδοθεί ε, διαφέρουν όσον αφορά την ε, κάλυψή τους. Συγγνώμη, μάλλον πρέπει να πάμε πίσω μια διαφάνεια. Όσον αφορά τις αδυναμίες, θα ήθελα να τονίσω τέσσερις τομείς που έχει εντοπίσει η Ένωση την οποία εκπροσωπώ. Καταρχά. από πλευρά τη βιομηχανία θα πρέπει να κοιτάξουμε και πέρα από τα σύνορα μα και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο ε, του καθεστώτο των μεταφορών στο γενικότερο και ευρύτερο διεθνέ ε, επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν ένα σύστημα ελέγχου των ε, μεταφορών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και προ την κατεύθυνση αυτή πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν ε, μεταρρυθμίσει στην οδηγία και στο σύστημα εξαγωγών και ότι όλο αυτό το σύνολο θα δημιουργήσει ένα στεναρό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη τι διεθνεί υποχρεώσει. Και επίση θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν με έξυπνο τρόπο, με ε, δέοντα σεβασμό προ την διαδικασία. Κατά δεύτερον, κάτι εξακολουθούν να ε, δίνουν υπερβολική έμφαση στον περιορισμό των εξαγωγών. Και κατά τρίτον, η διαδικασία πιστοποίηση είναι βαριά και για τι επιχειρήσει και για τι αρχέ που αξιολογούν κατά πόσον πληρούνται τα πρότυπα από τι επιχειρήσει. Και επίσης ε, υπάρχει η αίσθηση ότι είναι διαφορετικό το επίπεδο των ε, ε, ελέγχων στην διαδικασία πιστοποίησης και θα πρέπει να υπάρχει μια γενική επισκόπηση των συστημάτων και στα άλλα κράτη-μέλη όπου γίνεται η προμήθεια. Γιατί αν <coughs> υπάρχει σημαντική καθυστέρηση από τη... σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές για την παροχή τέτοιων αδειών, δεν υπάρχει ανάγκη να κοιτάξουμε τις διαδικασίες και τις δυνατότητες πιστοποίησης. Και τέλος, οι επιχειρήσεις, οι οποίες κυρίως έχουν έδρα σε διάφορα κράτη-μέλη, σε κάποιες περιπτώσεις ε, βλέπουν να είναι διαφορετικές οι του τι είναι μεταφορά προϊόντων και αυτό είναι σημαντικό. Και υπάρχει και έλλειψη συνένεση του τι σημαίνουν ε, ειδική κατασκευή, ειδικό σχεδιασμό για στρατηγική σχέση. Σε ό,τι αφορά, ε, σε ό,τι αφορά τώρα τι στρατηγικέ εξελίξει, ε, απομακρυνθήκαμε από την πλήρη ε, εξάρτηση από τις άδειε για τη χρήση τέτοιων ε, αδειών. εισαγωγή δε γενικών και καθολικών άδειων οδήγησε τα κράτη-μέλη να κάτσουν να σκεφτούν το τι αποτελεί ευαίσθητο και μη ευαίσθητο αντικείμενο. Και έτσι εξετάζουν το πώς θα πρέπει να γίνεται η αδειοδότηση για τα, τις δύο κατηγορίες ε, προϊόντων. Και τέλος, ε, οι πιστοποιημένες εταιρείε ε, και τα σχετικά σχέδια πιστοποιημένων εταιρείων έχουν φέρει στο επίκεντρο τη σημασία της συμβατότητας ελέγχου εξαγωγών και έτσι οι κυβερνήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ότι γίνονται κατανοητές στις σχετικές προδιαγραφές. Τέλος, θα ήθελα να κοιτάξω κάποιες από τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο σύστημα. Καταρχάς, η βιομηχανία πιστεύει ότι οι μεταφορές στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να υπόκειται σε ε, προδιαγραφές ε, αδειοδότησης ε, λιγότερο ευνοϊκές από ότι αυτές που χρησιμοποιούνται στη ΣΥΠΑ για εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν είναι σε μια ελεκτική θέση η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία σε σχέση με την, Ευρωπαϊκή, με την Αμερικανική διαδικασία ελέγχου αδειοδότησης. Επίσης χρειάζεται κοινή ερμηνεία των όρων και κυρίως του όρου specially designed, ειδικά σχεδιασμένου. Στη ΣΥΠΑ καταθέσουν δικούς τους ορισμούς και αυτό έχει ευρύες συνέπειες και σε ό,τι αφορά την διαδικασία διαδότησης και πολλά τέτοια αντικείμενα θα έπρεπε και πάλι να διαδοτούνται για να εξαγάγονται στο ιστορικό ή στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός όμως ότι δεν υπάρχει κοινό ορισμός οδηγεί σε διαφωνία μεταξύ των αρχών και γι' αυτό λοιπόν τα κρατημέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν επί κοινών ορισμών στα πλαίσια της συμφωνίας του Βασενάρ σε ό,τι αφορά ε, τα, την εξαγωγή τέτοιων αντικειμένων. Και αν δεν το καταφέρουμε, τουλάχιστον να υπάρχει ένα συμβατός ορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον ΕΙΠΑ. Θέλουμε να υπάρχει λοιπόν εναρμονισμένη διαδικασία και θα πρέπει να ακολουθείται και ένας κοινό μορφότυπος ό,τι αφορά τους όρους χρήσης και επίση θα πρέπει να ωφελούνται τα προϊόντα αυτά από το καθεστώς ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ζητούμε να μην υπάρχουν επιπλέον προδιαγραφές για την επαναεξαγωγή ούτε για τα αντικείμενα ούτε για τα εξαρτήματα τα οποία εξαγάγουν ε, οι εταιρείε, οι πιστοποιημένε εταιρείε. Και τέλο, τι αφορά τι πιστοποιημένε εταιρείε, πιστεύουμε ότι το σχέδιο πιστοποιημένων εταιρείων δεν λειτουργεί όσο έχει σήμερα και θα πρέπει να περάσει από αναθεώρηση για να είναι λιγότερο ε, βαρύ και να είναι πιο εναρμονισμένο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που εφαρμόζει σε όλες τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη μεταφορά προϊόντων στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λέμε γιατί πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις άμυνας θα πρέπει να έχουν εύρωστα προγράμματα που θα αποτυπώνουν ε, και τα προϊόντα και το εύρωστο την κάμα των προϊόντων τους, αλλά και την περιπλοκότητα της σύνθεσής τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σίλβες Τσάλβερς. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η παρουσίασή σας και ξεκάθαρα και τα αιτήματά σας και κατάλαβα ότι εκπροσωπείτε το σύνολο των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στον αμυντικό τομέα. Θα δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Πέλτς, η οποία συγκράτησε πολλά από τις δύο τελευταίες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σημειώσω το πόσο ενδιαφέρουσες ήταν ε, οι δύο παρουσιάσεις. Άκουσα προσεκτικά τα αιτήματα και τις ανησυχίες των εκπροσώπων της βιομηχανίας. Εμείς θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν σήμερα προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τα γραφειοκρατικά βάρη, να μειώσουμε τα γραφειοκρατικά βάρη καλύτερα και να δημιουργήσουμε ένα πεδίο θα έλεγα δίκαιο και ισότιμο για το σύνολο των κρατών μελών ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα επιπλέον μέσο το οποίο θα έχουμε στη διάθεσή μας αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Όπως είπαν οι ομιλητές, υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις για τη χρήση του μέσου και έχουμε νομίζω κάποιες δυνατότητες βελτίωσης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τη σημασία που έχει η διαδικασία πιστοποιήσεων των επιχειρήσεων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι επιχειρήσεις ε, θα έλεγα ε, θα το σκέπτονται πριν ξεκινήσουν μια τέτοια διαδικασία. Τα πλεονεκτήματα δεν είναι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή αν ε, υπερβαίνουν τις περιπλοκές. Συνεπώς λοιπόν απαιτείται η διαδικασία να διευκρινιστεί καλύτερα. Τα μέσα ε, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι πάρα πολλά λόγω των οικονομικών περιορισμών και γι' αυτό οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης όχι μόνο άμεσα στον αμυντικό τομέα αλλά γενικότερα στην καθημερινή δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να διευκρινιστούν κάποια σημεία τα οποία όπως είπα έχουν σημασία να διακρίνουμε ανάμεσα σε ευαίσθητα και λιγότερο ευαίσθητα προγράμματα και προϊόντα. Σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λοιπόν αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα ήταν καλό όλες οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη οδηγία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές στα κράτη-μέλη μεταξύ τους και αυτές οι διαφορές πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει πάντως να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο ότι δαπανώνται πάρα πολλά χρήματα, ευρωπαϊκά κεφάλαια και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε σχέση με την Αμερικανική βιομηχανία σε μειονεκτική θέση. Ε, κάποιος από τους ομιλητές αναφέρθηκε ε, στα, στη μεγάλη σημασία που έχουν εδώ οι ορισμοί και οι συγκεκριμένες κατηγορίες των προϊόντων. Είναι σημαντικό εδώ να υπάρξει πρόοδος. Λοιπόν, ευχαριστώ τους ομιλητές. Θα μου δώσανε ε, όπλα, θα έλεγα, για την επόμενη μου έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά δεν μπορώ να επιδείξω τέτοιε γνώσεις όσο οι προλαλήσαντε. ωστόσο θα ήθελα όσον αφορά τι δύο τελευταίες ομιλίε, ε, να θέσω μια ερώτηση. Ο εκπρόσωπος ε, του Φιλανδικού Υπουργείου Αμήνη ε, πολύ σωστά είπε ότι δεν μπορούμε πολύ απλά να πούμε ότι η προστασία των εθνικών συμφερόντων αποτελεί εμπόδιο για την εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η τελευταία ομιλία του εκπροσώπου της ε, EASD μας δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια αγορά με εθνικά εμπόδια τα οποία δεν ε, σχετίζονται απαραίτητα με ε, πολιτικά στοχευμένα μέτρα, αλλά έχουν να κάνουν με παραδόσεις ε, εντός των διαφόρων χωρών. Για παράδειγμα, η χώρα μου δυσκολεύεται πολύ κατά την εξαγωγή, διστάζει μάλλον ε, να εξάγει αμυντικό υλικό, παρότι συμμετέχει στην εσωτερική αγορά. Και έτσι πολλά από τα πλεονεκτήματα που ανέφερε ε, ο Γάλλος εκπρόσωπος μετριάζονται. διότι η Γερμανία ζητάει προέγκριση σχετικά με την ε, χρήση των προϊόντων αυτών σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο της ε, Γαλλίας ε, αλλά και του εκπροσώπου του βιομηχανικού τομέα. Να ρωτήσω, υπάρχουν προβλήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η ευρωπαϊκή πολιτική συγκεκριμένα ώστε να πετύχουμε συνέργειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, οι κατακαιρματισμένες εθνικές αγορές ε, να γίνουν μια ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και θα ξαναδώσω το λόγο στους δύο πανελίσεις. γιατί τους ετέθησαν ερωτήσεις και θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση. Μιας και πρόκειται για ένα διάλογο μεταξύ του Τσάλιβερς και που ήθελε μια ενιαία ερμηνεία του Special Designed ως όρο και του κυρίου Καρλιέ ο οποίος ε, μίλησε για το επίπεδο της Γαλλίας ε, σε κατά πόσον το Special Designed αυτό στη Γαλλία συνάδει με την αρχή και τον ορισμό των άλλων χωρών. Θα μπορούσατε λοιπόν να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα σας παρακαλώ και στις ερωτήσεις που έθεσαν του τους Σα Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και για να επανέλθω στα σημεία αυτά που σχολιάσατε. για τη διαπίστωση της σχετική με την εφαρμογή της οδηγίας. Ίσως τα μέσα να είναι παρόντα, αλλά ίσως και να μην χρησιμοποιούνται με εναρμονισμένο τρόπο. Συμφωνούμε με αυτό. Όπως βλέπετε προσπαθούμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να καθορίσουμε κάποιους κοινούς καταλόγους στρατιωτικού υλικού και καταλόγους χωρών προς τις οποίες μπορούμε να επανεξάγουμε. Αυτά θα έλεγα θα δώσουν ε, ουσία στα μέσα τα οποία ε, μας παρέχει η οδηγία αν δεν έχουμε τα μέσα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις προβλέψεις. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή. Σχετικά τώρα με τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε για την ενιαία αγορά προϊόντων άμυνας ή αμυντικού υλικού καλύτερα, στον τομέα της ολοκλήρωσης των βιομηχανιών υπάρχει το θέμα των μέσων που χρησιμοποιούνται και των αδειών εξαγωγής. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ολοκλήρωσης, αν θέλετε, ε, μεγάλων βιομηχανιών ανάμεσα στην Kraus Maffei και στην Nexter ε, υπήρξε μια σημαντική υποστήριξη της γαλλικής κυβέρνησης και της γερμανικής κυβέρνησης για αυτήν την επανένωση, συγχώνευση ή συνεργασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σωστή πολιτική και εδώ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συνεργασία στον τομέα των βλημάτων ή πυράβλων ανάμεσα <coughs> στην Ένωση και σε άλλες χώρες όπως η Ρωσία προσπαθούμε να καταλήξουμε σε εναρμονισμένες λίστες. Είναι ένα παράδειγμα περαιτέρω εναρμόνισης, παράδειγμα των, της χρήσης των μέσων που επιτρέπει η οδηγία. Μιλήσαμε για τις ατομικές αδειοδοτήσεις, οι γενικές αδειοδοτήσεις και οι σφαιρικές αδειοδοτήσεις είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην Γερμανία και επιτρέπει να ορίσουμε ένα σύνολο προϊόντων στρατιωτικών που μπορούν να εξαχθούν και στα πλαίσια ε, προγραμμάτων συνεργασίας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στα πλαίσια ε, μιας ε, βιομηχανικής συνεργασίας. Τώρα για την τελευταία ερώτηση για το Specially Design for Military Use. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει ε, μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Αυτό έγινε με μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους Γερμανούς. Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε ε, για να βρούμε μια μέθοδο η οποία να χρησιμοποιείται με απλό τρόπο από τους βιομηχάνους. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στις ιδέες που έχουν εκφράσει οι Αμερικανοί και για να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο Τσίλβερς, δεν νομίζω ότι θα έχουμε δυσκολίες για να δούμε μαζί με τους Αμερικανούς πώς θα εφαρμόσουμε από τη μία μια ευρωπαϊκή αν θέλετε αντίληψη και από την άλλη να είναι συμβατή και να εφαρμόζεται παράλληλα με την αντίστοιχη των Αμερικανών η ερμηνεία που δίνουμε είναι παρόμοια. Αλλά δεν έχουμε τους καταλόγους που ταυτίζονται. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αμερικανική αντίληψη. Να πω πάντως προς τον κύριο Τσίλβερς ότι υπάρχει τρόπος χρήσης των καταλόγων αυτών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές απόψεων ε, μεταξύ μας όσον αφορά το από πού ξεκινήσαμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Ε, αυτό με καθησυχάζει. Επιτρέψτε μου ε, επίσης να αναφερθώ στο θέμα των εμποδίων. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές όπως είπε και ο Γάλλος συνάδελφος. Εάν εξετάσουμε το, την βιομηχανία στην Ευρώπη και κατακαιρματίσουμε μια εταιρεία και έχουμε διάφορους κλάδους σε διάφορα κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχουμε τρόπο αδειοδότησης ώστε η συνεργασία να πραγματοποιείται ομαλά και να λειτουργεί η εταιρεία εξίσου αποτελεσματικά με το εάν λειτουργούσε εντός ενός κράτους μέλους, διότι αλλιώ υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν θέλαμε να υπάρχουν. Με καθησυχάζει λοιπόν το ότι εξετάζεται πολύ προσεκτικά τα προβλήματα αυτά. Γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα της ε, MDBA και της συνεργασίας ε, μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης με καθησυχάζει το θέμα του ειδικού σχεδιασμού. Επίσης με καθησυχάζει το γεγονός ότι πραγματοποιείται ε, δουλειά μεταξύ των κρατών μελών για τη βελτίωση της εφαρμογής, ότι εξετάζονται τα ευαίσθητα και μη ευαίσθητα προϊόντα και έχει γίνει πολλή δουλειά τον τελευταίο χρόνο περίπου ε, πάνω σε μια σειρά θεμάτων. Όσον αφορά την διαδικασία πιστοποίησης, επιτρέψτε μου να επανέλθω σε αυτήν. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ε, θα εξελιχθούν οι συζητήσεις και να συνεργαστούμε στενά με όλους, ώστε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα ικανοποιήσει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει πραγματικά επικοδομητικός διάλογος μεταξύ των διαφόρων πλευρών ε, του ζητήματος αυτό. Και έτσι περνάμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα της ακρόασής μας ε, ό,τι αφορά τα θέματα τέτοια προϊόντων άμυνας και θα δώσω το λόγο Και θα ήθελα να δώσω λοιπόν το λόγο σε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για την ευρωπαϊκή διάσταση των, ε, του θέματο γιατί η κυρία Τάνσα Γιακολά είναι ε, επικεφαλής ε, του European Synergies και Innovation και ε, επικεφαλή ε, της στρατηγικής για τη βιομηχανία και των ευρύτερων ευρωπαϊκών πολιτικών. Και θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε τυχαίος είναι ο αντίκτυπος της ρυθμίσης της εσωτερικής αγοράς σε ό,τι αφορά γενικότερα τις δυνατότητες ε, του κλάδου της άμυνας. Ευχαριστώ πολύ και για το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε να έρθω να μιλήσω στην Επιτροπή σας σήμερα. Επιτρέψτε μου καταρχάς ε, να σας θυμίσω το προφανές, ε, γιατί χρειαζόμαστε μια ανοιχτή αγορά ε, πιο αγορά αμυντικών προϊόντων πιο διαφανή. Δεν θα λειτουργήσει καλά εάν δεν υπάρχει μια καλή διαφανής αγορά, η οποία πρέπει να έχει διάφορες διαστάσεις. Καταρχάς έχουμε την νομική διάσταση και ενώ τις δύο οδηγίες που διέπουν τη λειτουργία της αμυντικής αγοράς, το θέμα δηλαδή της συζήτησης μας σήμερα. Δεύτερον, έχουμε την πολιτική διάσταση της αγοράς αυτής. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε ότι η αγορά αμυντικού εξοπλισμού δεν είναι αποκλειστικά εμπορικό θέμα, έχει συχνά πολιτικές ε, και στρατηγικές προεκτάσεις για τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, η ασφάλεια προμήθειας είναι πολύ σημαντική ε, στο θέμα αυτό. Γι' αυτό οι αγορές προϊόντων αμήνης ε, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι αγοράζει κανείς, αλλά και από ποιον. Τρίτον, έχουμε και την επιχειρησιακή διάσταση προμήθεια αμυντικών ε, προϊόντων ε, συνδέεται με την ασφάλεια της Ευρώπης ε, και, τους πολίτες, και των πολιτών της. Και αυτό είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την προμήθεια αμυντικού υλικού. Ο τίτλος της παρέμβασής μου συνδέεται με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και έχει να κάνει με την εφαρμογή και την χρήση που γίνεται των οδηγιών και αναφέρομαι στις ε, οδηγίες ε, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών στον τομέα της άμυνας ε, και για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων θεωμένων με τον τομέα της άμυνας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η λειτουργία και ο αντίκτυπος των οδηγιών. Όπως υπόθηκε, ετοιμάζονται οι σχετικές μεταρρυθμίσεις και αναμένονται εντός του 2016 στο Κοινοβούλιο. Και βέβαια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις. Να θέσω λοιπόν κάποια θέματα ε, τα οποία έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη μας όσον αφορά ε, την ε, οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών στον τομέα της άμυνας. Οι συζητήσεις μας με εμπειρογνώμανους των κρατών μελών έχουν οδηγήσει το εξή. Καταρχάς, οι δημόσιες συμβάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οδηγίας είναι τόσο λίγες διότι είδαμε σημαντική μείωση ε, των συμβάσεων ε, γενικά. Χαιρόμαστε που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει σημειωθεί η πρόοδος ε, και βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση μακροπρόθεσμα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή της οδηγίας. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις που δημιουργούν κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, για την υπεργολαβία φαίνεται να δημιουργούνται προβλήματα όσον αφορά τον στόχο των διατάξεων αυτών, που είναι να διευκολύνουν ε, την ε, διασυνοριακή πρόσβαση, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει στενά το θέμα αυτό για παράδειγμα μέσω της συμβουλευτικής ομάδας για την πρόσβαση στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου είμαστε και εμείς παρατηρητές. Ε, τρίτον, ε, ο αριθμός των διασυνοριακών ε, συμβάσεων στο πλαίσιο της οδηγίας. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερες αναλύσεις για να καταλάβουμε τους λόγους ε, για τους οποίους ε, είναι περιορισμένες ε, οι συμβάσεις αυτές και περιμένουμε και τη σχετική έκθεση της Κομισιόν για να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Και τέταρτον, όπως ήδη είπε ο κύριος καθηγητής, ίσως είναι πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε συμπεράσματα διότι γενικά απαιτούνται 5 με 10 χρόνια για την πλήρη εφαρμογή και χρήση μιας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει ήδη κάνει μια πρώτη αξιολόγηση σχετικά με την ε, οδηγία για τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Ε, το αποτέλεσμα της πρώτης αυτής αξιολόγησης, το οποίο έχουμε ε, δημοσιεύσει και στα κράτη-μέλη μας, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο άμεσο εμπόδιο στην συνεργασία που να απορρέει από την οδηγία. Η μη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όχι όμως, δεν οφείλεται όμως συγκεκριμένα στην οδηγία. Λίγα λόγια για το μέλλον. Όπως είπα νωρίτερα, ε, ο βασικός ε, στόχος ε, των δημοσίων συμβάσεων είναι να παρέχονται συστήματα και προϊόντα τα οποία χρειάζονται για να διασφαλίσουν την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αλλαγές στο περιβάλλον όσον αφορά την ασφάλεια και τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, μας αναγκάζουν να εξετάσουμε με διαφορετικό μάτι το μέσο που υιοθετήθηκε το 2009 εξετάσουμε εάν μας ε, παρέχει αυτά που χρειάζονται στον ε, σημερινό κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα. Επίσης, ε, όσον αφορά τις πιθανές βελτιώσεις, έχουμε την κλασική οδηγία και την οδηγία στους κοινοβουλευτικούς οργανισμούς που μπορούν να μας εμπνεύσουν όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας. Επίσης, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην δεύτερη οδηγία της δέσμης μέτρων αυτών ε, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεδομένων με τον τομέα της άμυνας ε, είναι κάτι που αφορά κυρίως ε, τα Υπουργεία ε, Αμήνης, αλλά όχι μόνο, μπορεί να σχετίζεται και με τα Υπουργεία ε, Εμπορίας, Εμπορίου και Εξωτερικών. Η ασφάλεια προμηθειών είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό η καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ε, μπορεί να ε, συμβάλλει στην αύξηση της ε, ασφάλειας προμηθειών εντός της Ευρώπης και μπορούμε έτσι να έχουμε καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Θέλουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια προμήθεια εντό τη Ευρώπη και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα παρακολουθεί στενά τι εξελίξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη σήμερα συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των ερευνών της ε, Κομισιόν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσθέσω ή να επαναλάβω τίποτα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας αυτής και ε, δεν, έχει, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα τις δυνατότητες της οδηγίας. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν διαφορετικέ προϋποθέσεις ε, όσον αφορά τις άδειες μεταφοράς προϊόντων. Με την ανάλυση της κατάστασης θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα των θεμάτων αυτών. Στόχος είναι να έχουμε εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εθνική εφαρμογή της οδηγίας αυτής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γενικές άδειε για μεταφορές προϊόντων. Όπως είπα νωρίτερα, το επόμενο ορόσημο θα είναι οι ε, ε, εκθέσεις εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι διατεθειμένος να στηρίξει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτών, ε, σεβόμενοι απολύτω τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του καθενός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή ήταν η σύντομη παρέμβασή μου στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μιλήσατε γρήγορα, αλλά όλοι καταλάβαμε το μήνυμά σας. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Πέλτς να σας απαντήσει ίσως και να κάνει και τις γενικές παρατηρήσεις για τις ομιλίες που προηγήθηκαν. Φτάνουμε στο τέλος του hearing. Ας κάνει λοιπόν παρατηρήσεις για το σύνολο των ομιλιών που προηγήθησαν. Ευχαριστώ και πάλι, Πέτρα. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους τελευταίους πανελίστες. Οι δημόσιε συμβάσει σε προϊόντα αμήνη είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να γίνει σαφή ρύθμιση. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ξεκάθαροι οι κανόνες μας είναι ουσιώδου σημασία αυτή για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλου του ε, φορεί. Πρώτου καταλήξω στα τελικά μου, καταρρεκτικά μου σχόλια, θα ήθελα να θέσω και μία ερώτηση. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκεκριμένα μέτρα για τις αρχές δημοσίων συμβάσεων που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς ακόμα και σε περιπτώσεις διοργάνωσης κοινών διαγωνισμών. Και εγώ πάντα είχα την εντύπωση ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο της οδηγίας, ε, καθώς ε, ισχύει για διάφορα στοιχεία, για διάφορους τομείς. Συμφωνώ απόλυτα ότι τα κράτη-μέλη θα, να κάνουν ό,τι περνάει το χέρι τους για να αξιοποιήσουν ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις οικονομίες κλίμακας και πραγματικά να χρησιμοποιήσουν την κοινή αγοραστή και τους δύναμη. Ωστόσο, και εδώ είναι το ερώτημα που έχω να θέσω, τα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια υπήρξε κάποιο προηγούμενο κοινή διοργάνωση διαγωνισμού θα ήθελα καταρχάς ε, να ακούσω την απάντηση στην ερώτηση αυτή, πρωτού προβώ στα καταληκτικά μου σχόλια, Πρόεδρε. Θέσατε λοιπόν μια ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε λοιπόν να απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Και θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η κυρία αναγκάστηκε να φύγει, είχε άλλε υποχρεώσει. σω όμω υπάρχει κάποιο άλλο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να απαντήσει στο όνομά τη. Θα μπορούσατε λοιπόν να απαντήσετε σε την τελευταία ερώτηση της κυρίας Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστώ. Είμαι ο επικεφαλής ε, υπεύθυνο του τμήματος για την ε, οδηγία αυτή. Έχουμε κάποια παραδείγματα, ίσως όχι τόσο ξεκάθαρα, αλλά για προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν από κοινού από κάποια κρατημέλη, αλλά πραγματικά είναι περιορισμένα τα παραδείγματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική αξιολόγηση. Είμαστε στη φάση συλλογής δεδομένων, αλλά πραγματικά σε ό,τι αφορά του κοινού διαγωνισμού εξακολουθούν να αποτελούν ένα πρόβλημα. Δεν βλέπουμε τέτοια κοινή χρήση των διατάξεων της οδηγίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εξαίρεση στην οδηγία που επιτρέπει στα κρατη να αναπτύξουν α, τέτοια προϊόντα στον τομέα της άμυνας. Έχουμε κάποια παραδείγματα κοινών ε, έργων ανάπτυξης, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι η οδηγία αυτή εξακολουθεί να είναι αρκετά ουδέτερη. Δεν βλέπουμε λοιπόν τέτοια τεράστια ανάπτυξη του δυναμικού αυτού σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά του ε, πέντε επιρρογνώμονες μα, οι οποίοι ήλθαν από τι ε, διαφορετικέ άκρε τη Ευρώπη για να μα μιλήσουν για το θέμα αυτό. Μήπω κάποιο από εσά ή κάποιοι από εσά, ε, θα ήθελα να πάρουν το λόγο για μισό λεπτό για να κάνουν κάποιο σχόλιο. Αν το επιθυμείτε να σας δώσω το λόγο, αν όχι, φυσικά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αν θέλετε βέβαια κάτι οπωσδήποτε να εκφράσετε στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, ε, μην διστάσετε να σηκώσετε το χέρι και να ζητήσετε το λόγο. Όχι, ήσασταν πειθαρχημένοι, δεν επιθυμείτε το λόγο και μιλήσατε εντό των χρονικών ορίων. Θα ήθελα λοιπόν να σα ευχαριστήσω εκ νέου και δεν πρόκειται να προβώ στην εξαγωγή ιδιαίτερων ε, συμπερασμάτων. Να εκφράσω μερικέ σκέψει όμω. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η ενιαία αγορά και οι απαιτήσει του τομέα της άμυνας είναι δύο ψυχές που δεν συνδυάζονται τόσο εύκολα απαραίτητα και εκ παραλλήλου θεωρώ ότι όλοι είμαστε πεπισμένοι να συγκεράσουμε αυτές τις διαφορετικές ε, ανάγκες και δεν πρόκειται μάλιστα για μια απαραίτητη ασυμβατότητα υπάρχει κάποια δυσκολία αλλά δεν υπάρχουν ασυμβατότητες ε, απόλυτες. Είμαστε λοιπόν στο, εν το μέσο μιας διαδικασίας ακολουθούμε μια πορεία και σε κάποιες περιπτώσεις, ε, ξέρετε, η πορεία είναι πιο σημαντική από την επίτευξη του τελικού στόχου. Όταν ε, μιλάμε για την ενιαία αγορά, σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Μα ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η ενιαία αγορά. Πάντα θα προχωρά, θα εξελίσσεται. Και υπάρχει και κάτι παραπλανητικό στην ίδια την έννοια της ολοκλήρωσης της ενίας αγορές. Ένα παράδειγμα επιπρόσθετο σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που καταβάλουμε για να λειτουργεί καλύτερα η εσωτερική αγορά. Προφανώς πρόκειται για ένα σημαντικό κλάδο, ένα κλάδο τον οποίο θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Αλλά νομίζω ότι κλείνουμε τη σημερινή ακρόαση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι προφανώς ο... δεν κινηθήκαν όλα όσο γρήγορα θα επιθυμούσαμε, θα ευχόμαστε και αυτό φαίνεται και στην έκταση αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Επόμενη εβδομάδα. αλλά σαφώ υπάρχει πρόοδο και θεωρώ ότι συχνά τονίστηκε και στα αγγλικά το κατά πόσο χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή, προσαρμογή χωρίς όμως να προδώσουμε την ίδια τη φιλοσοφία και την ιδεολογία της ενιαίας αγοράς. Ακόμα και αν δεν είμαστε πιστοί στο γράμμα του νόμου. Όλα τα ζητήματα που είναι ζητήματα άμυνας προφανώς ε, ε σχετίζονται με τον πυρήνα της ιστορικής ε, και γεωγραφικής παράδοσης των κρατών μελών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό από το μέγεθος της χώρας της ίδιας. Υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες οι οποίες έχουν ε, ιδιαίτερη παράδοση σε ό,τι αφορά την ε, ε, βιομηχανία της άμυνας και είναι πραγματικά ε, μεγάλη η παράδοση τους αυτή και άλλα κρατημένα δεν έχουν την ίδια ιστορία και παράδοση και θα πρέπει προφανώς να προσεγγίσουν αυτές οι ιστορικές πραγματικότητες καθώς και οι γεωγραφικές πραγματικότητες που διαφέρουν στην Ευρώπη και στην ιστορική αγορά και θεωρώ ότι ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας ε, αυτό είναι σημαντικό γιατί πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητος. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα λοιπόν. Έχουμε μπροστά μας αρκετά θέματα. Βλέπουμε ότι η έννοια της άμυνας, η ίδια η έννοια της άμυνας, δεν είναι μόνο εξωτερική άμυνα, αλλά υπάρχει εδώ και ένα στοιχείο εσωτερικής άμυνας απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι σε αυτά τα δράματα τα οποία χτύπησαν τις πρωτεύουσές μας εδώ και λίγες εβδομάδες, ακόμα και τη δική μας πρωτεύουσα εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εργαστούμε και στα πλαίσια της εσωτερικής άμυνας. Αυτό δικαιολογεί και απαιτεί να υπάρξει μια συνεργασία καλύτερη. Ο εχθρός είναι κάποιος ο οποίος είναι απολύτως κοινός και όχι μόνο είναι κοινό ο εχθρό, αλλά κυκλοφορεί στο εσωτερικό του σύνορων μα Και είναι πραγματικά προσαρμόσιμο στι διαφορετικέ καταστάσει. En de défense intérieure également sur euh, χαμελέον ο εχθρό τρομοκράτη προσαρμόζεται στι διαφορετικέ συνθήκε και γι' αυτό απαιτείται να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις αρχές καταστολής, στις ένοπλες δυνάμεις κτλ. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα επί του οποίου απαιτείται χρόνος, απαιτείται αυτός ο χρόνος προσαρμογής να χρησιμοποιηθεί με χρήσιμο τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιμείνει ε, προς την κατεύθυνση αυτή και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει η διαδικασία αυτή που είναι μια δύσκολη διαδικασία να συνεχιστεί χωρίς να χάσουμε τον στόχο που έχουμε μπροστά μας, να μην ξεχάσουμε και τα στάδια από τα οποία θα πρέπει να περάσουμε, να συνεχίσουμε δηλαδή να ακολουθούμε την πορεία που έχουμε ήδη χαράξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλειωσε λοιπόν το hearing για την άμυνα. Κυρία Γκαλπέλτ, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ίσως να ευχαριστήσετε και εσείς τους προσκεκλημένους μας και στην συνέχεια αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε στις 5 Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για λίγα λεπτά λοιπόν, αμέσως μετά την, κατα... την παρέμβαση εν κατακλείδη της κυρίας Πέλτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά συνοψίσατε το βασικό μήνυμα αυτής της ακρόασης. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπατε δεν θα μπορούσα να τα είχα πει πιο καθαρά από ό,τι τα είπατε εσείς. Δεν απομένουν λοιπόν πολλά να πω, πέρα από το να ευχαριστήσω τους ομιλητές, τους προσκεκλημένους μας, για την σημαντική συμβολή τους, τις σημαντικές προτάσεις τους. Δεν ε, θέλω να επαναλαμβάνομαι κι εγώ, διότι ήδη πήρα το λόγο. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις μόνο να κάνω, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει τα σωστά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το πόσο έχουν προχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε την ταχύτητα πρόοδου μας. Δεύτερον, οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά άμυνας θα πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζονται, να συνεχίσουμε να τις αναλύουμε και μόνο αφού αναλύσουμε την κατάσταση να υποβάλουμε νέες προτάσεις. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε να νομοθετήσουμε. Είναι πολύ ιδιαίτερη αγορά, η αγορά προϊόντων αμήνης. Ήταν πάντα κατακαιρματισμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για να μειώσει τον κατακαιρματισμό, αλλά όπως είπε πολύ σωστά ο Πρόεδρος, έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα μέχρι να μπορούμε να μιλάμε για ενοποιημένη αγορά μείνεις στην Ευρώπη. να αναφερθώ σε κάποιους τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. οι επιμέρους συμβάσεις, τα προγράμματα συνεργασίας και συγκεκριμένοι αποκλεισμοί οι οποίοι μπορούν να στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά τι θα κάνουμε για όλα αυτά στο μέλλον. Όλα αυτά δεν αποτελούν αναποσπαστό μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς ε, προϊόντων αμήνης και απαιτείται να γίνουν αλλαγές. Πάντως έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει πολύ στενό περιθώριο ευελιξίας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συμβαίνει αυτό. Κάποιοι λόγοι είναι ε, πιο σωστοί από κάποιους άλλους. Πολλά κράτη-μέλη προσπαθούν να ευνοήσουν τη δική τους ε, βιομηχανία άμυνας. Τα κράτη-μέλη διστάζουν να πούνε σε τέτοιες σχέσεις αμοιβαίας εξάρτησης και γι' αυτό δεν εκμεταλλεύονται τις συνέργειες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στις κινήσεις μας και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Άμυνας ε, θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξος. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες επίσης όσον, όσον αφορά την ε, οικονομία κλίμακας. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως όμως ε, σας είπα θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την ευρωπαϊκή αγορά και να αναλύσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και πάλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας. Ε, μας έδωσαν πολύ τροφή για σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, Έφτασε η ώρα Πέντε. Εγκαίρως λοιπόν ξεκινάμε το δεύτερο τμήμα της συνάντησής μας σήμερα το απόγευμα. Η ΙΜΚΟ είχε ζητήσει να υπάρξει μία μελέτη για την προσπάθεια καταμέτρησης του κόστους του μη Σέγγεν γνωρίζουμε όλοι και βλέπουμε με πόνο πολλοί από εμά να κλείνουν πάλι τα σύνορα, ελπίζουμε προσωρινά σε ορισμένες περιπτώσεις, στο εσωτερικό της Ένωσης, στα εσωτερικά σύνορα, ίσως τελικά να είναι σε αμφισβήτηση ένα τμήμα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αλλά εδώ δεν κάνουμε μια γενική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από αυτά τα θέματα. Βρισκόμαστε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και είναι θεμητό για μας να αναρωτηθούμε αν κάτι τέτοιο θα βλάψει την εσωτερική αγορά. Το ξέρουμε αυτό, αλλά με ποιο τρόπο και ποια θα είναι η εμβέλεια της βλάβης. Ζητήθηκε αντίστοιχα κάτι από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για θέματα πιο νομικά και για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Εμείς όμως ασχολούμεθα με την κυκλοφορία των αγαθών και των προϊόντων που μειώνουν την δυναμική της εσωτερικής αγοράς. Θα ακούσουμε μία παρουσίαση λοιπόν των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ θα έχουμε την δυνατότητα να σχολιάσουμε και να θέσουμε ερωτήσεις. Η τελική μορφή της μελέτης αυτής δεν θα είναι διαθέσιμη παρά στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια τα οποία προβλέπονται για το κόστος του μη Σέγγεν ξεκινούν από μια κατάσταση ελέγχου της ε, καθημερινότητας ε, σε μια ακραία κατάσταση της πλήρους αποκατάστασης των εσωτερικών συνόρων. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ μαζί μας και θέλω μάλιστα να ευχαριστήσω Ε, τον δόκτορα Ματίας Λούκε, ο οποίος είναι εξωτερικός εμπειρογνώμων της Επιτροπής μας. Θα του δώσω το λόγο σε λίγα λεπτά. Είναι σύνιορ ερευνητής του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία και καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου για τη Διεθνή Οικονομία. Θα δώσω επίσης το λόγο στην κυρία Στριτ Βόρομ, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Εργάζεται στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου στην υπηρεσία έρευνας και τεκμηρίωσης. Δεν ξέρω με ποια σειρά θα μιλήσετε, αλλά αν σας ικανοποιεί η σειρά την οποία ε, ήδη έχω δώσει, έχει το λόγο ο κύριος Σωματίας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλησπέρα σε όλους, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα στην παρουσίαση αυτή να αναφέρω την δουλειά που έκανα με τον Τιμπρή από το Λόρβαν σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία του πώς γίνονται ε, η αξιολόγηση του κόστους του μη Σέγγεν και μετά να σας αναφέρω και τι συμπεράσματα, σε τι συμπεράσματα έχουν καταλήξει και άλλες μελέτες που έχουν γίνει για να δούμε ε, συνολικά πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε το κόστος του Μισέγγερ και τέλος ε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό, πώς μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να επανέλθουν σε ένα πλήρες καθεστώς Σέγγεν δεδομένου και του κόστους και ποια είναι τα ενδεχόμενα ωφέλη τα οποία θα μπορούσαν να υπολογίσουν τα κράτη-μέλη να περάσουμε κατευθείαν στην ουσία στο ψητό, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Η μεθοδολογία λοιπόν περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Καταρχάς ε, διαπιστώνουμε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι επιβάλλουν κάποιο κόστος στον κόσμο και καθυστέρηση. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε πώς αυξάνεται το κόστος του διεθνούς εμπορίου ως αποτέλεσμα των ε, ελέγχων αυτών στα σύνορα και των ελέγχων ε, οχημάτων ενδεχομένω. Αυτό είναι σε πρώτη φάση λοιπόν ο υπολογισμός της αύξησης του κόστους και κατά δεύτερον όταν ε, βρούμε ποια είναι το επιπρόσθετο κόστος των συνοριακών ελέγχων τότε μπορούμε να αναρωτηθούμε το ε, σε τι αντιστοιχεί αυτό σε κόστος επιπλέον για τον καταναλωτή. Πώς επηρεάζει αυτό το πραγματικό εισόδημα του καταναλωτή. Αυτά λοιπόν είναι δύο διαφορετικά βήματα. Να μιλήσω καταρχάς για το πρώτο βήμα, γιατί εδώ υπάρχει, πρέπει να σας πούμε ότι πολλές έρευνες υπολογίζουν το κόστος ε, του συνοριακών ελέγχων σε σχέση με το εμπόριο απλά προσθέτοντας μερικά στοιχεία. κοιτάμε δηλαδή πόσα φορτηγά περιμένουν στα σύνορα, για πόσο χρονικό διάστημα, υπολογίζουμε πόσο κοστίζει το χρονικό διάστημα και τα προσθέτουμε όλα αυτά. Αυτή είναι μία μέθοδος. Μία άλλη μέθοδος είναι να αναρωτηθούμε κατά πόσον αυτό τα περιλαμβάνει όλα ή μήπως ε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα πρέπει να προσθέσουμε, τον αντίκτυπο του Σέγγεν στο διμερές εμπόριο στην ε, Ευρώπη σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία. Να δούμε δηλαδή κατά πόσον αυξήθηκε το διμερές εμπόριο μεταξύ των μελών λόγω του Σέγγεν και να το υπολογίσουμε αυτό και να έχουμε και μια εναλλακτική, εναλλακτικό υπολογισμό της αύξησης του κόστους ε, του διεθνούς εμπορίου λόγω των συνοριακών ελέγχων. Το δεύτερο βήμα της ανάλυσης είναι λιγότερο σημαντικό, γιατί εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των διάφορων μοντέλων που χρησιμοποιούνται για να μεταφραστεί η αύξηση του κόστους σε αύξηση κόστου για τον καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν ε, μπορούμε να είμαστε αρκετά σύντομοι. Α περάσουμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο και να δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε υπολογισμού ε, βάσει τη πρώτη μεθόδου, από κάτω προ τα πάνω ένα α σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση στα σύνορα. Δεν μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία στον πίνακα, αλλά αυτό που θα μπορείτε να βρείτε ενδεχομένω είναι ότι Έχουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επικεφαλίδες στις στήλε και στην αριστερή πλευρά του πίνακα και ο πίνακας αναφέρει πόσα φορτηγά περνούν ε, τα σύνορα του κάθε κρατούς μέλους. Τους ίδιους πίνακες καταρτήσαμε και για λεωφορεία, πούλμαν και ιδιωτικά οχήματα και στη συνέχεια κάνουμε και κάποιες εναλλακτικές εικασίε για το χρονικό διάστημα το οποίο θα χρειάζεται να περιμένουν τα οχήματα στα σύνορα, σε κάθε σύνορο, αν υπάρχουν και έρευνες των οχημάτων. Και εδώ μιλάμε 10, για 10-20 λεπτά ανά αυτοκίνητα και 30 έως 60 λεπτά για φορτηγά και λεωφορεία. Και υπάρχουν και διαφορετικές τιμές για το πόσο θα χρειαστεί να περιμένει ένα όχημα. Και το πόσο κοστίζει η αναμονή. Και αυτό φυσικά εξαρτάται από τι κάνετε αυτοκίνητα, αν κινείται για επαγγελματικού σκοπού ή για σκοπού αναψυχή. Εδώ φυσικά υπάρχουν διαφορέ. Στην επόμενη διαφάνεια τα προσθέτουμε όλα αυτά, όλα τα κόστη σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Και πάλι σε κάθε στήλη έχουμε τη χώρα που επιβάλλει τους ελέγχους. Αυτό είναι αρκετά καινοτομικός μέθοδος, γιατί ξέρουμε και ποιες χώρες επιβαρύνονται με το κόστος η πρώτη χώρα είναι ασφαλώς η Αυστρία. Η πρώτη λοιπόν στήλη υποδεικνύει ποιο θα ήταν το κόστος αν η Αυστρία επέβαλε πλήρη συνοριακό έλεγχο σε, όλες, σε όλα τα σύνορα. Συνολικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και προκύπτει ότι και η ίδια η Αυστρία θα επιφανεθεί μόνο με 100 εκατομμύρια του κόστους αυτούς, ενώ μεγάλο ποσοστό θα επιβαρύνει την Γερμανία και την Ιταλία. Φυσικά επειδή είναι ε, χώρα διέλευσης η Αυστρία, πολλά φορτηγά περνούν από την Αυστρία. Και έτσι νομίζω ότι με πολύ επικοδομητικό <coughs> τρόπο προβάλλεται το κόστος όπως κατανέμεται στις διάφορες χώρες. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που βλέπω τέτοια ε, κατανομή και χαίρομαι που το TNL το έκανε αυτό. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα της μεθοδολογίας 1α, της απλής δηλαδή, του απλού αθροίσματος των, της ώρας αναμονής στα σύνορα. Υπάρχει και το συνολικό άθροισμα και το συνολικό άθροισμα λοιπόν του κόστους το βλέπετε κάτω δεξιά. 5 δις ευρώ το συνολικό κόστος ενδεχόμενης πλήρους επιβολής νοριακών ελέγχων από όλα τα κράτη-μέλη. Πέντε της το έτος. Το ενδοκινητικό εμπόριο ανέρχεται στα 3.000 δις το έτος. Το ΑΕΠ ε, ε, Ευρώπης, το στολικό ΑΕΠ της Ευρώπης είναι 12.000 ε, δις ανά Είναι πολύ μικρό το ποσό δηλαδή συγκριτικά. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί. Ε, αυτό είναι όλο. Αρκεί να κοιτούμε τον μέσο χρόνο αναμονής του οχήματος και αυτό να αποτελεί τη βάση του υπολογισμού του κόστους. Όχι, όχι, γιατί ενδεχομένως, ε, αν ξέρω ότι θα χρειαστεί να περιμένω μισή ώρα, να μην βγω καν στον δρόμο. και ενδεχομένω άμα ξέρω ότι θα πρέπει να κολλήσω δύο ώρες στην κίνηση μπορεί και να μετακομίσω. Και φυσικά αυτό έχει άλλε συνέπειε. και το ίδιο συμβαίνει ασφαλώ και για τι υπηρεσίε μεταφορά με φορτηγά γιατί πρέπει να κάνουν το πρόγραμμά τους, να βγάλουν πίνακε για την φορτωσή και εκφόρτωση. Αν ξέρουν λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι θα υπάρχει καθυστέρηση, όλα αυτά επηρεάζονται με τη σειρά τους και το κόστος μπορεί να σχετίζεται και κυρίως με την αβεβαιότητα για τη διάρκεια της καθυστέρησης και όχι με την ίδια την καθυστέρηση και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντική η μέθοδος 1β όπου ο κόσμος εξετάζει ποιος είναι ο αντίκτυπος του Σέγγεν, ιστορικός πώς ε, στο διμερές εμπόριο και τι θα επηρεαστεί ως αποτέλεσμα του παγώματος του Σέγγεν. Και να δούμε στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν τα αποτελέσματα. Να εστιαστούμε στην ε, μελέτη Φέμπερ από το Ίδρυμα του Μονάχου που είναι πολύ προσεκτική και διαπιστώνει η έρευνα ότι για κάθε έλεγχο Σέγγεν που περιλαμβάνεται σε διμερές επίπεδο, ε, μάλλον για κάθε σύνορο ιστορικά, η αύξηση του εμπορίου με το Σέγγεν ήταν 2,7%. Για τη Γαλλία και τη Γερμανία θα περιμέναμε για παράδειγμα αύξηση 2,7% του εμπορίου μεταξύ Πορτογαλίας και Πολωνίας επειδή πρέπει να περάσει τέσσερα σύνορα το ενδεχόμενο προϊόν, η αύξηση ήταν τέσσερις φορές 2,7%. Και επίσης, πόσο μειώθηκε το κόστος του εμπορίου α, για ως αποτέλεσμα της επιβολής του Σέγγεν. Και βλέπουμε στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν ποιο είναι το ποσό αυτό. Εδώ έχουμε διάφορες εικασίες σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα του εμπορίου και το πώς τα εμπόδια στο εμπόριο επηρεάζουν το διμερές εμπόριο. Και βλέπετε ότι η αύξηση είναι μεταξύ 0,4 και 0,9% μάλλον η αύξηση του κόστους ανά σύνορο μπορεί να υπολογιστεί μεταξύ 0,4 και 0,9% για τα εμπορευόμενα αγαθά και το ίδιο για τις υπηρεσίες που α, ε, αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, όπου ο αντίκτυπος είναι και λίγο πιο μεγάλος. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο, η επιβολή ελέγχων του, στα σύνορα πριν το Σέγγεν θα αύξανε το κόστος του εμπορίου κατά τουλάχιστον 0,4% και ενδεχομένως και πιο πολύ για κάθε σύνορο που διασκίσετε. Και αυτό ασφαλώς είναι πολύ παραπάνω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως, τα οποία ενδεχομένως να αντιπροσωπεύουν 0,1% της αξίας του εμπορίου. Άρα η αύξηση του κόστους είναι πολύ παραπάνω από αυτό που θα υποδείκνυε η πρώτη αυτή μέθοδος 1α. Το επόμενο ζήτημα που ανακύπτει είναι ασφαλώς ε, το πώς λειτουργεί αυτό και τι αποτέλεσμα έχει αυτό για τον καταναλωτή. Κάποια αγαθά προφανώς καθίστανται πιο αγαθά, άλλα ενδεχομένως να φθηναίνουν γιατί οι εξαγωγείς προτιμούν να πουλούν εσωτερικά στην Εμεδαπή. Και κάποια εγχώρια προϊόντα ενδεχομένω να παράγονται πιο πολύ σε πιο μεγάλε ποσότητε στην Ημεδαπή. Πολλά λοιπόν θα άλλαζαν και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο τη οικονομία, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά αντικειμενικοί. Και αν κοιτάξετε στην προηγούμενη διαφάνεια. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το ποια σύνορα υποθέτουμε ότι θα επηρεαστούν από τον έλεγχο των σύνοριακών. Τα κράτη-μέλη που εφήρμοσαν τέτοιους ελέγχους δεν καλύπτουν όλα τα σύνορα. Σε περίπτωση της Γερμανίας, για παράδειγμα, ε, οι έλεγχοι αφορούν συγκεκριμένα τα σύνορα με την Αυστρία, με την Αυστρία με τη Σλοβενία, ίσως και με την Ιταλία στο μέλλον. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Άρα να προσέξουμε στο σημείο αυτό. Και ίσω το πιο σχετικό σενάριο είναι το σενάριο υπαριθμών 3, όπω ονομάζεται, όπου η ιδέα είναι η εξή ότι οι χώρε θα εφαρμόσουν ε, ελέγχου στι μεγάλε μεταναστευτικέ οδού. Ε, από τα Βαλκάνια προς την Βορειά Ευρώπη. Και έτσι το κόστος σε ό,τι αφορά το πραγματικό εισόδημα είναι κάτω από το 0,1% ό,τι μέθοδος υπολογισμού και να εφαρμόσουμε. Και αυτό ισχύει και για τη Γερμανία και για την Αυστρία. Άρα και πάλι το κόστος, αν ρεαλιστικά υποθέσουμε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε περιορισμένες ε, σε περιορισμένα τμήματα των συνόρων που υπάρχει συγκεκριμένη απειλή, τότε το κόστος είναι περιορισμένο ποσοστό. Αν όλοι εφαρμόσουν ε, ελέγχου σε όλα τα σύνορα, βλέπετε ότι είμαστε στο δεύτερο τέο σενάριο, το 0,4% αύξηση κόστου, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό. Άρα, ε, όλα εξαρτώνται από το ποιο είναι ο στόχο των χωρών αναφορικά με τους νεριακούς έλεγχους. Αν υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη του ΣΕΓΕΝ, το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι μια στοχευμένη διεξαγωγή ελέγχου στα σύνορα. Και έτσι περνάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Προφανώ υπάρχει κόστο. Μπορεί να μην είναι τεράστιο, όπω δείχνουν οι έρευνε, μπορεί να μην είναι τεράστιο. Άρα το μεγάλο θέμα είναι γιατί το εφαρμόζουν αυτό το σύστημα οι χώρε αν θέλουμε να εφαρμόσουμε και πάλι πλήρως τους κανόνες του Σέγγεν. Κάποιες χώρες ε, θέτουν το θέμα της ασφάλειας, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο μετά τις τρομοκρατικές ε, επιθέσεις. Άλλες ε, χώρες, όπως οι σκανδιναβικές, λένε ότι δεν μπορούν να έρχονται ανεξέλεκτα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στη χώρα μας. Άρα κάπως πρέπει να αντιδράσουμε. Στην περίπτωση της Γερμανίας, νομίζω ότι προσφάτως που μίλησα με ένα αξιωματούχο τη κυβέρνηση μου εξήγησε ότι δεν ε, επιστρέφουμε του πρόσφυγε όποιο θέλει να ζητήσει άσυλο στην Γερμανία θα εξετάσουμε την άτησή του. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα εκατομμύριο ε, ανθρώπου όπω το 2015. Πρόκειται για θέμα ασφάλεια, πρόκειται για θέμα αστυνόμευση. και έτσι θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν την κατάσταση. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι όλοι, αν θέλουμε όλοι να επανέλθουν στην κατάσταση που προβλέπει το ΣΕΝΓΕΝ, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα εξωτερικά σύνορα. Όταν θα υπάρξει πλήρη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων, τότε θα είμαστε ασφαλείς πλέον και οι χώρες θα μπορούν να επανέλθουν στους κανόνες του Σένιον πλήρως. Και τέλος να πω και δύο λόγια για το τι μπορούμε να κάνουμε στο έντο μεταξύ. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της πλήρους και κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνάρων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Πολλοί έλεγχοι γίνονται με πολύ πρόχειρο τρόπο. Και αυτό ασφαλώς αποστέλνει και ένα μήνυμα, αλλά γιατί όταν οι χώρες δεν ε, δημιουργούν ειδικέ υποδομές, αυτό δίνει την εντύπωση ότι θα είναι κάτι προσωρινό. Αλλά από την άλλη, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη και κάποια υποδομή, ενδεχομένω τα πράγματα θα πάνε πιο γρήγορα. Αν ε, χρειάζονται λοιπόν αυτή η έλεγχοι επί προσωρινή βάση, τουλάχιστον να υπάρχει και μια κατάλληλη υποδομή για να υπάρχει μια ελάχιστη περίοδο αναμονή. Και στην τελική ανάλυση προφανώς θα πρέπει να υποστηριχθούν οι χώρες εκείνες όπου θα πρέπει να γίνει η εξωτερική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, οι περιφερειακές χώρες, γιατί δεν μπορούν να φέρουν μόνες τους την ευθύνη της υποδοχής των προσφύγων και της επεξεργασίας της διεκπαιρέωσης των αιτήσεων για άσυλο. Θα πρέπει λοιπόν με συνεκτικό τρόπο να ασφαλιστούν τα εξωτερικά σύνορα και αυτό αποτελεί ευθύνη όλων των συμμετεχόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λούκε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Βόρουμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε την έκθεσή μας για το κόστος του μη Σέγγεν και για τις επιπτώσεις της αποκατάστασης των ελέγχων στα σύνορα. και τις επιπτώσεις που θα έχει σε οικονομικό επίπεδο η αποκατάσταση του ελέγχου των συνόρων στην εσωτερική ενιαία αγορά. Πρέπει να δούμε καταρχάς ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας εσωτερικής αγοράς η Συμφωνία Σέγγεν συμπληρώνει τις τέσσερις βασικές ελευθερίες του άρθρου 26 της Συνθήκης. Διευκολύνει λοιπόν τις εμπορικές ροές και βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μια μελέτη που αφορά και το 16 μας δίδει εμπειρικά στοιχεία αυτής της προστιθέμενης αξίας. Εδώ βλέπουμε ότι σε πολλούς τομείς, σε επίπεδο ΑΕΠ, σε επίπεδο εσωτερικού εμπορίου, κινητικότητας, υπάρχουν μετρήσιμα πλεονεκτήματα για την ύπαρξη αυτής της ενιαίας αγοράς. Οι τέσσερις ελευθερίες επιτρέπουν τη σωστή κατανομή των πόρων και έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, υψηλή παραγωγικότητα, και ευρύτερες αγορές που επιτρέπουν οικονομίες κλίμακας. Σήμερα οι ελευθερίες αυτές αμφισβητούνται μέσω της εισαγωγής ελέγχων. Ακόμα και σε προσωρινό επίπεδο αυτό δημιουργεί προβλήματα στις διασυνοριακές ροές. Ποιες θα είναι οι πραγματικές επιπτώσεις λοιπόν. Θα σε τρεις φάσεις. Καταρχάς, ο έλεγχος θα προκαλέσει άμεσο κόστος, θα υπονομεύσει τα πλεονεκτήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια και δεν θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Θα φυγούν οι πολίτες, θα φυγούν οι επιχειρήσεις. Αυτό θα επηρέασει και άλλους τομείς στη συνέχεια με σημαντικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με την μελέτη τέσσερις τομείς θα επηρεαστούν. Πρώτον, η, αγορά αυτών οι οποίοι εργάζονται σε μεθοριακές περιοχές, είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι, θα αυξηθεί ο χρόνος εργασίας τους και οι αγορές αυτές θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές. Δεύτερον, λόγω της απώλειας χρόνου στα σύνορα θα υπάρξει μείωση στα ταξίδια για αναψυχή και στον τουρισμό. Αυτό θα οδηγήσει σε μια πολυδιάσπαση και της διαδικασίας θεωρήσεων και αυτό θα οδηγήσει σε επιπλέον απώλειες. Και τέλος υπάρχει το θέμα της εμπορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ε, μεγαλύτερη αναμονή για τους οδηγούς φορτηγών θα δημιουργήσει αύξηση του κόστους του προσωπικού, καθυστέρηση της παράδοσης των προϊόντων. Πέρα από τον ίδιο τον τομέα των μεταφορών, θα υπάρξουν επιπτώσεις και στο μέγεθος του εμπορίου και στο επίπεδο των τιμών που θα αυξηθούν και αυτό θα οδηγήσει σε χαμηλότερη κατανάλωση και αυτό θα επηρεώσει φυσικά, θα επηρεάσει συγγνώμη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Ε, ένας ε, ε, μακροπρόθεσμος τομέας είναι η απόδοση των ομολόγων. Αν οι αγορές εγκαταλείψουν τον Σέγγεν, αυτό θα επηρεάσει και τις χρηματαγορές αρνητικά. Κάποιες χώρες θα θεωρείται ότι δεν ανήκουν πλέον στον πυρήνα τον ευρωπαϊκό και η απόδοση των κυβερνητικών κρατικών ομολόγων θα αυξηθούν για χώρες που θα θεωρηθούν αυτόματα πιο επικίνδυνες χώρες ε, σε οικονομικό επίπεδο. Αν η τιμή λοιπόν, το τίμημα αυξηθεί, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και σε επίπεδο ε, επιτοκίων και αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για την πραγματική οικονομία στο σύνολό της. Να δούμε τώρα τα αποτελέσματα της έρευνας πιο αναλυτικά. Δύο βασικά σενάρια μια κατάργηση, μια επιβολή μάλλον για δύο χρόνια των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ή μία αορίστου χρόνου κατάργηση της συμφωνίας του Σέγγεν. Υπάρχουν δύο δυνατότητες και εδώ. Η, κατάργηση να αφορά συγκεκριμένες χώρες, 7 προς το παρόν, ή να αφορά το σύνολο των χωρών. Υπάρχει φυσικά το θέμα του κόστους του μη Σέγγεν. Κάθε χώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κόστος της αποκατάστασης των ελέγχων στα σύνορα. Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι αυτό σημαίνει 70 ευρώ κατά κεφαλήν επιπλέον. Αυτό μας οδηγεί σε 7,1 δις συνολικά για τις 7 χώρες επαναλαμβάνω. Υπάρχουν και άλλα σενάρια, όπως είπα, καταρχάς μετά από δύο χρόνια και για λίγες χώρες, δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, γιατί ακούσαμε κάποιες λεπτομέρειες, θα επηρεαστούν άμεσα οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι διαμεθοριακοί εργαζόμενοι, θα επηρεαστούν οι μετακινούμενοι για λόγους αναψυχής και τουρισμού, θα επηρεαστούν επίσης οι μεταφορές προϊόντων. Ανάμεσα στις 7 χώρες η Αυστρία είναι αυτή η οποία θα φύγει περισσότερο λόγω της διαμετακόμισης προϊόντων και λόγω του υψηλού αριθμού των διαμεθοριακών εργαζομένων. Μετά από δύο χρόνια το κόστος θα δημιουργήσει καθυστερήσεις και οι καθυστερήσεις επιπλέον κόστος και θα επηρεαστεί και η τουριστική όπως είπα δραστηριότητα. Αυτό θα φτάσει τα 5 δις σε δύο χρόνια για τις έξι χώρες μέλη. Για τη δεύτερη περίπτωση, δύο χρόνια κατάργηση για όλες τις χώρες. Οι ίδιοι τομείς θα επηρεαστούν, 1,7 ε, εκατομμύρια διαμεθοριακοί εργαζόμενοι, αύξηση του χρόνου μετακίνησης κατά 50 περίπου λεπτά την ημέρα, αυτό θα οδηγήσει σε υψηλές οικονομικές απώλειες. Ο τουρισμός επίσης θα επηρεαστεί και αυτό θα επηρεάσει φυσικά όλα τα κράτη-μέλη. Θα επηρεαστούν επίσης ε, και οι εμπορευματικές μεταφορές και θα φτάσουμε σε 3,6 δις σε ετήσια βάση. Για το σύνολο λοιπόν, για δύο χρόνια κατάργηση για όλες τις χώρες, θα φτάσει τα 51 δις συνολικά, από 26 μάλλον μέχρι 51, για όλες τις χώρες, για δύο χρόνια. Να δούμε τώρα το σενάριο της πλήρους κατάργησης του Σέγγεν για 10 χρόνια, για να έχουμε μία μακροπρόθεσμη προοπτική θα υπάρξουν κάποιες ευρύτερες μακροοικονομικές αλλοιώσεις. Καταρχάς, αν μιλήσουμε για, τον περιορισμένο αριθμό χωρών που καταργούν το Σέγγεν, οι χρηματαγορές θα το ερμηνεύσουν σαν μήνυμα ότι οι χώρες αυτές δεν επιθυμούν να ανήκουν στον ευρωπαϊκό πυρήνα. Η απόδοση των κρατικών ομολόγων θα αυξηθεί και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κρίσεις, αποσταθεροποιήσεις και αυτό θα οδηγήσει ε, ε, και τις πιθανότητες ε, αποτυχίας των συγκεκριμένων οικονομιών και αδυναμίας πληρωμής χρέους. και οι χώρες αυτές θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για τα χρέη τα οποία επιστρέφουν. Και θα υπάρξει φυσικά εξ αυτού και μείωση των ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν λιγότερες επενδύσεις και αύξηση των επιτοκίων και αρνητική, ε, αρνητική επιρροή στους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Τώρα, ε, για μια πιο μακρά περίοδο έχουμε πάλι δύο σενάρια. Πρώτον έχουμε την επίπτωση για το ΑΕΠ στις 7 χώρες, αυτό σημαίνει 70 δις ζημία. Και ταυτόχρονα αν υπάρξει και μια ευρύτερη κρίση, οι χώρες αυτές θα πρέπει να προβλέψουν και άλλα 170 εκατομμύρια σε επίπεδο ε, δημοσιονομικού κόστους. Τώρα για μια πλήρη διακοπή της λειτουργίας του Σέγγεν μετά από 10 χρόνια το κόστος ε, θα προκληθεί κυρίως από την ε, αρνητική επιρροή στις εμπορικές συναλλαγές, στον τουρισμό και στους διασυνοριακούς εργαζομένους. Αυτό θα επηρεάσει το σύνολο του εσωτερικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επηρεάσει την ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας. Αν υπάρξει μια πλήρης διακοπή της ισχύω του Σέγγεν, αυτό θα ερμηνευθεί από τους επενδυτές σαν ένα βήμα προς τα πίσω για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι μια καλή για επενδύσεις περιοχή όπως ήταν στο παρελθόν. Αυτό θα επηρεάσει τις χρηματικές ροές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, μία πλήρης κατάργηση ε, σε αόριστο χρόνο, για αόριστο χρόνο του Σέγγεν, θα οδηγήσει σε μία απώλεια του ΑΕΠ σε ετήσια βάση κατά 0,14%. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε απώλειες 230 δις σε δεκαετή βάση στην περίπτωση που είναι περιορισμένες οι χώρες που εγκαταλείπουν το Σέγγεν, βλέπετε στον πίνακα τον προηγούμενο, συμπερασματικά να πω ότι η συμφωνία του Σέγγεν θεωρείται ένα σημαντικό συμπλήρωμα της ενιαίας αγοράς που διευκολύνει την ενδοκινοτική εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και σε επίπεδο ελεύθερης διακίνησης. Οι μελέτες δείχνουν ότι το κόστος της κατάργησης της ελεύθερης διακίνησης είναι σημαντικό, ίσως όχι τόσο σημαντικό όσο πίστευαν ορισμένοι. Αλλά οι επιπτώσεις δεν θα είναι οι ίδιες σε όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες θα επηρεαστούν, αλλά άλλες περισσότερο από ότι ε, κάποιες υπόλοιπες. Συμπερασματικά λοιπόν για το σύνολο της περιοχής Σέγγεν το συνολικό κόστος υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 51 δις για μια διακοπή διετή και τα 230 δις σε δεκαετή βάση για πλήρη κατάργηση. Ε, μια τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι Υπάρχουν και τα έμεσα κόστη τα οποία δεν είναι εύκολο να μορφοποιήσει κανείς, σαν παράδειγμα η απώλεια εμπιστοσύνη στο ευρώ. Αυτό είναι κάτι που θα βλάψει συνολικά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ε, γιατί το Σέγγεν είναι ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Να σας ζητήσουμε συγγνώμη γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο για τη μελέτη αυτή απαιτούνται περισσότερες μελέτες για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις εφόσον υπάρχει ο επαρκής χρόνος. Και εφόσον το επιθυμείτε σαν ΙΜΚΟ, η υπηρεσία EPRS του Κοινοβουλίου μπορεί να συνεχίσει τις αξιολογήσεις της για το κόστος του μη Σέγγεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μας. Ήμουν οικονομολόγος, είμαι οικονομολόγος, κατανοώ τις μεθοδολογικές δυσκολίες που είχατε να αντιμετωπίσετε. Ο κύριος Σβάμπ. Ο κύριος Κοέλιο, παρακαλώ. I want to thank the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ερευνητές για τη μελέτη αυτή. Και θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Δεν έχω ερωτήσεις, παρατηρήσεις έχω, τρεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξής. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα. Πριν χρόνια εξετάσαμε το κόστος ε, έλλειψης της Ευρώπης ε, για να αιτιολογήσουμε την πολιτική της ενιαίας αγοράς που αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Γνωρίζαμε τότε ότι η ελεύθερη κινητικότητα αποτελεί κλειδί για την ευημερία της Ευρώπης. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα όσον αφορά το Σέγγεν, το κόστος αναστολής ε, της ζώνης Σέγγεν δείχνει ότι είχαμε δίκιο τότε που λέγαμε ότι χρειαζόμαστε ανοιχτή Ευρώπη. Και θα έπρεπε να καταλήξουμε και τώρα στο ίδιο συμπέρασμα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι φυσικά υπάρχει κόστος. Οι ομιλητές μίλησαν πολύ σωστά γι' αυτό. Υπάρχει το κόστος των νέων ελέγχων, το κόστος στα σύνορα, το κόστος που προέρχεται από τον αντίκτυπο στο εμπόριο, το κόστος απώλειας του χρόνου, το κόστος απώλειας του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, το κόστος από την απώλεια τουρισμού. Δεν υπάρχει λόγος Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα, υπερβολικά πολλά μέτρα προστασίας όμως, ε, μέτρα ασφάλειας, ε, συνεπάγονται αυξημένο κόστος. Από τη δική μας ε, πλευρά λοιπόν θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο θέμα ιδεολογικής θέσης, είμαστε υπέρ της Ευρώπης και υπέρ της ελεύθερης κινητικότητας, αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος. Έχουμε υπολογισμό του κόστους ε, αναστολής της ζώνης Σένιεν, ακρίβει υπολογισμό. Και θα ήθελα επίσης να πω, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, τα οικονομικά στοιχεία αυτά δεν είναι μόνο αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη, όπως είπαν άλλωστε και οι ερευνητές. Η καταστροφή της ζώνης Σέγγεν σίγουρα δεν αποτελεί λύση. Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσουμε, αλλά σίγουρα η λύση δεν είναι η καταστροφή της ζώνης Σέγγεν, διότι κινδυνεύουμε όχι μόνο να χάσουμε να καταστρέψουμε, όπως υπόθηκε πολύ σωστά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, αλλά κινδυνεύουμε να προσθέσουμε στην οικονομική κρίση που ήδη αντιμετωπίζουμε το κόστος ε, αναστολής ε, τη ζώνη Σέγγεν. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τη ζώνη Σέγγεν. Και τώρα έχουμε περισσότερα επιχειρήματα στο χέρι μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σουάπ, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για εσάς για την παρουσίαση που μας κάνατε για τις δύο αυτές ε, έρευνες και την αξιολόγηση μάλλον των άλλων ε, ερευνών και θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος Κάρλος Κουέλια από την Πορτογαλία. Νομίζω ότι με τα αριθμητικά στοιχεία αυτά μπορούμε να καταδείξουμε πόσο σημαντική είναι για την ευρωπαϊκή αγορά και τους ευρωπαίους πολίτες ε, η μη αναμονή στα πρώην σύνορα και ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο και το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναμονή, φυσικά συνδέεται και με κάποιο συγκεκριμένο κόστος, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί με μακροοικονομικό τρόπο και τη σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για τους πρόσφυγες έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το θέμα της ασφάλειας και αυτό θα πρέπει να επιληθεί, αλλά στη συζήτηση ήταν δύσκολο να ε, εντοπίσουμε ποιες δυνατότητες θα καταδικάζαμε σε θάνατο άμα επιβάλαμε τα εθνικά σύνορα. Και στην τελική ανάλυση πολλοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να λύσουμε το θέμα της ασφάλειας και της προσφυγικής ροής ε, κρατώντας τα σύνορα ανοιχτά. Γιατί όλοι τελικά έχουμε μεγάλο συμφέρον να μην είναι ανοιχτά τα εσωτερικά σύνορα για το εσωτερικό εμπόριο, αλλά φυσικά όλα τα κρατημέλη θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών σύνορων, για να μην έχουμε θέματα ασφάλειας. Άρα όλα αυτά είναι αλληλεσυνδεόμενα συνδεόμενα και γι' αυτό λοιπόν ήταν σημαντικό το γεγονός ότι έγινε μια διάμεση μελέτη όταν ξεκίνησε αυτή η έντονη συζήτηση και στην τελική ανάλυση τα ανεξάρτητα ιδρύματα στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία ε, μας ε, υπέβαλαν γρήγορα τα αριθμητικά αυτά στοιχεία και τους υπολογισμούς τους και σίγουρα θα είναι ε, πολύ επίκαιρο το πολιτικό ζήτημα για να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να προβάλλονται γρήγορα τα στοιχεία αυτά και θα πρέπει να μην δίνουμε την ευκαιρία να συγκεντρώνουν άλλη την προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις έρευνες αυτές, οι οποίες νομίζω ότι θα έχουν εμπρέπτες συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε, Ανδρέα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Και δεν ε, είναι και τόσοι βουλευτές που είναι εδώ να κάνω λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να θέσω ε, να κάνω διαφορά μεταξύ των επιστημονικών και πολιτικών ε, σκέψεων σε επίπεδο τεχνικό, επιστημονικό. Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Καταρχάς, όταν σκέφτομαι τα ζητήματα αυτά, Νομίζω ότι πάντα υπάρχει ένα αντίθετο αποτέλεσμα να λάβουμε υπόψη και έχει ενδιαφέρον. Το εμπόριο μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας και η Ευρώπης σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, τη μεταφορά μέσω φέρι, μέσω τούνελ και σε ό,τι αφορά και τη μεταφορά προς το Βέλγιο. Είναι σαφές ότι σε ένα μέρος όπου δεν ισχύει η ζώνη Σέγγεν και όπου υπάρχουν έλεγχοι, στα εμπορεύματα και στους ε, πολίτες και μάλιστα οι έλεγχοι αυτοί έχουν επιταθεί με την προσφυγική κρίση και όχι τόσο με την τρομοκρατική κρίση. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε ότι σε ό,τι αφορά την επανεισαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην ζώνη Σέγγεν, να δούμε τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη ζώνη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως που υπήρχαν πάντα τέτοιοι έλεγχοι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλη ροή, γιατί ξέρουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία παράγει μεγάλα, μεγάλα μηχανικών προϊόντων και σας μιλώ με τη, για τη σύνδεση με το Βέλγιο και τη Γαλλία, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, τέτοιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε και κάτι το οποίο θα θέσει υπό αμφισβήτηση τις εικασίες σας και τις ερευνές σας για το Σένιεν. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει πιο πολύ με τη μεθοδολογία. Θεωρώ ότι είναι μάλλον απίθανο να εγκαταλείψουμε πλήρως το Σένιεν η κατάσταση, το χειρότερο σενάριο είναι να παραμείνουν οι συμφωνίες μεταξύ των κρατών, μεταξύ των όμορων κρατών, αλλά δεν πρόκειται να επανεισαχθεί έτσι γρήγορα το σύστημα ελέγχου σε όλο το μήκος των συνόρων μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου. Για παράδειγμα έχουν επανεισαχθεί κάποιοι έλεγχοι και όσοι από εμά μετακινούνται πολύ μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας και τελειώνουμε ότι γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι κτλ. κτλ. Και καλό θα ήταν, θεωρώ, να το έχουμε και αυτό υπόψη για να δούμε τι θα σήμαινε αυτό ως εναλλακτική, πώς θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τα συντήματα. Και τώρα θα ήθελα να βάλω και αν θέλετε το πολιτικό μου καπέλα και να μιλήσω από την πολιτική μου ιδιότητα. Σε πολιτικό επίπεδο, στο τελική ανάλυση, η πρώτη αντίδραση όταν ακούμε τα στοιχεία αυτά είναι να σκεφτούμε ότι το κόστος είναι πολύ σημαντικό και παράλληλα με ένα κόστος το οποίο θα έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρρεύσει προς Θεού. Και νομίζω ότι ο κύριος Ματίας Λούκε το είπε στην αρχή ότι ενδεχομένως με το κόστος αυτό να φαίνεται πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι όσοι δηλώνουν ότι δεν θέλουν περισσότερη Ευρώπη θα μπορούσαν άντα να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτό το σενάριο σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θέμα εσωτερικής ασφάλειας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να θίξουμε και να θέσουμε το πολιτικό σκέλος του προβλήματος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που θα πρέπει να τονιστούν. Το πρώτο είναι αρκετά συγκεκριμένο. Το κόστος αυτό ε, ποιους τομείς θα επιβαρύνει στο σενάριό σας για τα 50 δισεκατομμύρια, για παράδειγμα, 200 δισεκατομμύρια. Υπάρχει κάποιος, ε, κάποιος κλάδος ο οποίος ε, παράγει 50 δισεκατομμύρια, γιατί το 50 δισεκατομμύρια μπορεί από μόνο του να μην σημαίνει κάτι. Αν λέγαμε, για παράδειγμα, ότι αυτά τα 50 δισεκατομμύρια αναλογούν σε όλο τον κλάδο ε, αναψυκτικών στην Ευρώπη, θεωρώ ότι τότε θα ήταν πολύ πιο ενδεικτικό το παράδειγμα. Και δεύτερη παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω. Και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε περισσότερο και ιδιαίτερα εμεί ω πολιτικοί και κυρίω εδώ στην Επιτροπή μα, στην Επιτροπή ε, Προστασία του Καταναλωτή. Ήταν το τελικό σα συμπέρασμα, αγαπητή κυρία θεωρώ ότι είναι θέμα φιλοσοφίας, νοοτροπίας, δυναμικής. Θεωρώ ότι το να επαναφέρουμε τα σύνορα, τους νοριακούς ελέγχους, θα έδινε ένα μήνυμα προς τις επιχειρήσεις. Ενώ όλοι μας έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ενωμένη, πιο ενοποιημένη, και μιλώ τώρα όχι ως πρόεδρος αλλά ως εκπρόσωπος της πολιτικής μου ομάδας. Είμαστε φεντεραλιστές, θέλουμε λοιπόν αυτή την αναμενή Ευρώπη. Και έτσι αυτό θα δημιουργούσε μια ελαστικότητα. Γιατί όταν δηλώνουμε τα σύνορα αυτό προφανώς αποτελεί κίνητρο και το αντίθετο ισχύει επίσης. Άρα, έχετε κάποια μοντέλα που θα μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε όλα αυτά, γιατί εγώ έχω αυτή τη βαθιά αίσθηση για να το θέσω διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για πολλά θέματα και διαρκώς ε, πραγματευόμαστε ε, ζητήματα όπως για παράδειγμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάποια περιοχή ε, Τη Ευρώπη που δηλώνουν ότι για παράδειγμα είναι δύσκολο να πωλήσουν τα προϊόντα του ε, σε κάποια ε, περιοχή τη Ευρώπη, γιατί δεν είναι ίδια τα δικαιώματα, το επίπεδο προστασία η συμπεριφορά του καταναλωτή και ούτω καθεξής. Μιλάμε για το ταχυδρομικό σύστημα, το κόστο και όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλέ ε, εταιρείε και μικρόμεσες επιχειρήσεις οι οποίες αποθαρρύνονται εκ των προτέρων και δεν κάνουν αυτό το βήμα για να επεκταθούν. Γιατί αποθαρρύνονται. Αποθαρρύνονται από όσους τους λένε ότι είναι διαφορετικοί οι καταναλωτές κτλ. Και θεωρώ ότι αν αύριο καταργούσαμε το Σέγγεν, θα δυσκολευόμασταν ακόμα περισσότερο να πείσουμε τις εταιρείες αυτές να επεκταθούν. Δεν είναι δηλαδή το θέμα μόνο το άμεσο κόστος. Τι θα γίνει... Επιπλέον αποθάρρυνση λοιπόν. Η εσωτερική αγορά είναι μια μάχη την οποία δίνουμε. Είναι ένας αγώνας, ένας πόλεμος. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις φοβίες, τους δισταγμούς, την αδάνεια. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε αυτές τις προσπάθειες, πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα και γι' αυτό πρέπει να τα θεωρήσετε αυτά τα ΟΗΠΑ σαν συμπληρωματικά στοιχεία, όχι σαν στοιχεία κριτικής σε αυτά τα οποία είπατε. Έχετε το λόγο για να κλείσετε αν θέλετε σε αυτά τα οποία είπαμε ε, ο κύριος Κοέλιο και εγώ, μιας και ο αγαπητός Ανδρέας αναχώρησε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας εκφράσω κάποιους συλλογισμούς μου για το θέμα αυτό. Ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις. Ξέρω ποιος είστε, αλλά μπορείτε να συστηθείτε. Ζήτω συγγνώμη, ναι, καταλαβαίνω. Άνδρου Λιόκελ από την ε, Europe Economics. Ε, έχω εξετάσει τις ποσοτικές στοιχείες της ε, έρευνας που μόλις παρουσιάστηκε. Θα εκφράσω κάποιες σκέψεις που γεννήθηκαν από τις παρατηρήσεις σας. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εμείς αναγνωρίζουμε στο εγγραφό μας ότι Φυσικά, οι χώρε ε, που επανεισάγουν τα σύνορα το κάνουν αυτό για συγκεκριμένο λόγο και πιστεύουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ωφέλη από αυτό. Δεν προσπαθήσαμε να ποσοτικοποιήσουμε τα ωφέλη που πιστεύουν ότι έχουν όσον αφορά την ασφάλεια κλπ δεν προσπαθήσαμε να συνδέσουμε οικονομικό όφελος με αυτά. Ε, εμείς επικεντρωθήκαμε στο κόστος αναστολής της ζώνης Σέγγεν και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν υποστηρίζουμε ότι αναλύσαμε αρκετά την κατάσταση ώστε να ισχυριζόμαστε ότι οι χώρες που ε, έχουν ε, εισάγει τα μέτρα αυτά το κάναν αυτό εις βάρος της ίδιας τους της οικονομίας. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι η ανάλυση μας δεν εξετάζει πολύ την κατανομή του κόστους. Για παράδειγμα, μέρος του δημοσιονομικού κόστους, καθότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που θα επηρεαστούν, έχει αυτή τη στιγμή πιστωτές ε, η Ελλάδα Δεν σημαίνουν όλα αυτά ότι θα πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια στα δάνεια τους, αλλά ότι θα υπάρχει ένα γενικότερο κόστος. Δεν έχουμε πει ποιος φέρει το επιπλέον κόστος που υπολογίσαμε. Επίσης θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες από τις άλλες προτάσεις που ακούστηκαν. Φυσικά θα ήταν χρήσιμο να έχουμε έρευνε για τι ε, συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις επανεισαγωγή των συνόρων, για παράδειγμα την αύξηση του χρόνου μεταφοράς κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο. Δεν είχαμε όμως πρόσβαση στα δεδομένα αυτά κατά τη ε, διαξαγωγή της έρευνας. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν νομίζω ότι θα αποτελεί καλό παράδειγμα, διότι εμείς επικεντρωθήκαμε κυρίως στα χερσαία σύνορα. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει επηρεαστεί, ε, έχει όμως πολλά θαλάσσια σύνορα, αλλά έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στα εσωτερικά χερσαία σύνορα. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν δεν θα μας ενδιαφέρει τόσο όσο άλλες από τις περιπτώσεις που εξετάσαμε. Επίσης ε, η ανάλυση ανατομέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ε, ποιοι τομείς επηρεάστηκαν από τις διάφορες μετακινήσεις και αυτό θα ήταν χρήσιμη διεύρυνση της έρευνάς μας. Μία ακόμα παρατήρηση έχω στην ανάλυση μας. Επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο πρώτο βήμα, όπως ε, ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτό να το παρατείνουμε, να εξετάσουμε και το έμεσο κόστος ε, στην ε, αλυσίδα προμήθειας, ε, διότι θα υπάρχουν δευτερογενείς συνέπειες αλλού. Για παράδειγμα, αν εγώ έχω περισσότερο χρόνο αναμονή στα σύνορα, μπορεί να αγοράζω λιγότερα προϊόντα. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τον τρόπο που διάφορες αντιδράσεις θα αυξήσουν το κόστος, διότι διάφοροι οικονομικοί παράγοντες ε, αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο απέναντι στη, στην αύξηση του κόστους διότι υποθέτουμε ότι ο κόσμο θα συνεχίσει να κάνει ακριβώ τα ίδια που κάνει τώρα, αλλά θα φέρει το αυξημένο κόστο. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ε, μέγιστη τιμή, διότι όλε οι προσαρμογέ που θα κάνουν θα μειώσουν το συνολικό κόστο. Βέβαια αυτό θα έχει μια άλλη σειρά πολύπλοκων συνεπειών, τις οποίε δεν είχαμε το χρόνο να εξετάσουμε. Έχει όμως ε, να κάνει με την όλη κατάσταση. Είχαμε περιορισμένο χρόνο. Σίγουρα δεν έχουμε αναλύσει επαρκώς την όλη κατάσταση, αλλά βρήκαμε διάφορα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια έχουν καταλήξει σε πολύ πιο υψηλά νούμερα, αλλά νομίζω κάπως ασυνήθιστο σε αυτά που κάναμε και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν θα πρέπει να πιστεύετε ότι η επανεισαγωγή συνόρων σε μέρος της ζώνης Σέγγεν δεν σημαίνει απλά μείωση του συνολικού κόστους. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει χειρό μήνυμα και ιδιαίτερα καθότι ε, αποστέλλεται το μήνυμα και όλα σε ότι κάποιες από τις εμπλεκόμενες χώρες δεν θα συνεχίσουν να είναι ε, μέλη της ζώνης Σέγγεν. Οι ε, συνέπειες όσον αφορά την ε, ιδιότητα με, κράτους μέλους της Ευρώπης για τις χώρες αυτές είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να εξετάσουμε ελαφρά την καρδία. Είναι το ερώτημά σας σχετικά με το ψυχολογικό κομμάτι και το έμεσο κόστος. Ε, αυτό δεν ήταν ε, στο πλαίσιο της αναφοράς της έρευνάς μας. Δεν μας το είχε ζητήσει. Αν θέλετε να το κάνουμε, τόσο το καλύτερο στη διάθεσή σας. Έχει σημασία αυτό, γιατί αυτό έχει σχέση με τη συμμετοχή στη ζώνη ευρώ και σε άλλα θέματα όπως οι πολιτιστικές αλλαγές και οι επιχειρήσεις δεν θα έρχονται στην Ευρώπη από τρίτες χώρες γιατί ήταν μια ανοιχτή αγορά ενώ τώρα τα πράγματα μπλέξανε. Ε, η αποκατάσταση των ελέγχων θα δημιουργήσει αρνητικά μηνύματα. Θα πω στους συντονιστές της ΣΥΜΚΟ την παρατήρησή σας γιατί πράγματι είναι κρίμα που το αίτημά μας δεν περιλαμβάνει. Θέλετε κάτι να πείτε? Εσείς όχι. Εντάξει, όσοι ήθελαν το λόγο το πήραν. Λοιπόν, θα ήθελα, εγώ όμως θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία άκουσα και τα οποία βρίσκω σημαντικά και δεν τα σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Δηλαδή οι διαφορές ανακράτως. Νομίζω ότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το ευρωπαϊκό, η το ευρωπαϊκό σχέδιο, η ευρωπαϊκή προοπτική είναι μια προοπτική αλληλεγγύης και στον οικονομικό τομέα και με πείσατε για το ότι το κόστος του Σέγγεν και αναφερθήκατε και στην Ελλάδα νομίζω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε ακριβώς την ιδέα αυτή για το κόστος του μη Σέγγεν γιατί έχουμε να κάνουμε με χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σήμερα, οικονομικές δυσκολίες, με προγράμματα αναδιοργάνωσης της οικονομίας τους. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα συμπεριληφθεί στην έρευνά σας, αλλά πρόκειται επίσης... Ε, αν υπάρξουν χώρες οι οποίες που καταργήσουν πλήρως το Σέγγεν. Και αυτό θα έχει ασφαλώς ε, και ε, σημαντικές ε, επιπτώσεις στο Σέγγεν. Δεν θα πρέπει λοιπόν το συνολικό κόστος ε, να αναιρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές και ότι ενδεχομένω να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης από κάποια χώρα. Όταν μίλησα πριν από λίγο για την Ηνωμένη Βασίλεια, γιατί το ανέφερα ως παράδειγμα. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ και ότι δεν είναι και στη ζώνη του Σέγγεν. Και δεν μιλάω για την πολιτική διάσταση, μιλάω για το οικονομικό σκέλος, την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία μάλλον που περνάει κρίση έχει ε, μεγάλους πόρους. Είναι, ε, έχουμε μεγάλο δυναμικό, είναι μεγάλη χώρα. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξη. Δεν είμαστε όλοι εξίσου ευάλωτοι και θεωρώ ότι η θέση αναμφισβήτηση του Σέγγεν θα για μια τέτοια διάκριση ε, των χωρών της Ευρώπης ε, και θεωρώ ότι και αυτό ως παράγοντας θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Bien. Euh, je pense que... Μάλιστα. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Ε, και συνάδελφοί σα, ε, οι οποίοι ε, μπορεί να μην προβλέπετε να πάρουν το λόγο, αλλά πήραν το λόγο και βοήθησαν στην κατάρτιση ε, έρευνα, πήραν το λόγο και σα ευχαριστώ λοιπόν όλου σα Σα ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή, Σα ευχαριστώ για την έρευνα, κατανοήσαμε καλά ότι θα έχουμε σύντομα και τα οριστικά αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία και προσμένουμε με μεγάλη αδημονία και κυρίως στη δική μας Επιτροπή αλλά και σε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι όντως οτιδήποτε αποτελεί τροχοπέδι στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των αγαθών ε, και οτιδήποτε αποδυναμώνει την ενιαία αγορά και το ευρωπαϊκό έργο δεν ναι. μπορεί παρά να βλάψει τους Ευρωπαίους και το οικονομικό σύστημα και τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ σας εύχομαι σε όλους. Αλλά συγγνώμη να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΜΚΟ θα λάβει χώρα στις 23 ε, ε, Μαΐου και στις 24 Μαΐου όλη την ημέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα με την πρόεδρο Βίκη Φόρτ, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί το απόγευμα γιατί είχε άλλε δοσμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.